As our uh, chairman is uh, not Κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος δεν θα είναι παρόν σήμερα και αύριο. Γι' αυτό θα αναλάβω εγώ την προεδρία της Επιτροπής αυτής, εγώ σήμερα και ο συνάδελφος κ. Κέρκοπ αύριο το απόγευμα. Αρχικά να σας ανακοινώσω ότι το σημείο 20 για την ε, συνεργασία διαχείρισης επιστροφής ε, σε τρίτες ε, χώρες και η πρακτική εφαρμογή της οδηγίας επιστροφής που προβλέπεται για αύριο έχει αναβληθεί. Αύριο το πρωί στις 9 θα αρχίσουμε τη συνεδρίαση συζητώντας το σημείο 10. για την Συμφωνία Πλαίσιο Ευρωπαϊκή Ένωση και Ινδονησία. Η κυρία Γκόμε, η συγγήτρια, ζήτησε να συζητηθεί αύριο το πρωί. Έπειτα θα συνεχίσουμε με το σημείο 9. Τρίτε χώρε, οι υπήκοοι των οποίων υπόκειται στην υποχρέωση θεώρηση για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων και τρίτε χώρε, οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή. Έπειτα, ψηφοφορία για το σημείο 10. 4. Δέσμευση και δίμευση των προϊόντων των εγκλήματο στην Ευρωπαϊκή Ένωση με συγκίτρια την κυρία Μακοβέη θα ψηφιστεί τελευταίο μετά από αίτημα τη συγκίτρια. Τώρα, οι διαπραγματεύσει για το πολιετέ συνομικό πλαίσιο και τι εσωτερικέ υποθέσει. Το σημείο, τα σημεία δηλαδή 15 και 18 της ημερήσιας διάταξης θα ολοκληρωθούν μεν, δεν θα προλάβουμε όμως να τα ολοκληρώσουμε αύριο. Γι' αυτό οι ψηφοφορίες θα αναβληθούν για τον Ιανουάριο του 2014. Και οι άλλες δύο εκθέσεις που έχουν σχέση με το δημοσιονομικό πλαίσιο, οι εκθέσεις Κολίνο και Μαρινέσκου, έχουν ολοκληρωθεί. Ωστόσο, η πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων εκδήλωσαν την επιθυμία να ψηφιστεί τον Ιανουάριο όλο το δημοσιονομικό πλαίσιο ως πακέτο μόλις ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για τον κανονισμό ορίζοντας. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για αυτές τις τροποποιήσεις, μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Δεν βλέπω αντιρρήσεις. Εγκρίνεται λοιπόν. Τώρα, έχω τη ε, συστάσει των συντονιστών προς έγκριση, ο εισηγητών. Εγώ, Κιν Καγκάλ, εισηγήτρια για την ΣΕΠΟΛ, την δημιουργία της ΣΕΠΟΛ, η κυρία Ρενάτε Βέμπερ για την απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τα συμπεράσματα του πολιτικού διαλόγου και της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών με την Κωνσταντίνα Ονδούρα Νικαράγουα Έπειτα, η κυρία θα είναι εισηγήτρια για την πρόταση κανονισμού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό για τον κατάλογο των τρίτων χωρών, κάτι και τον οποίο υπόκειται σε υποχρέωση θεώρησης. Και εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για τις συστάσεις αυτές των συντονιστών, μπορούμε να τις εγκρίνουμε. Δεν βλέπω αντιρρήσεις τότε. Επόμενη ανακοίνωση. Πέραν των προγραμματισμένων συνεδριάσεων της Επιτροπής ΛΥΜΠΑ έχουν προσθεθεί τρεις ακόμα συνεδριάσεις, στις 13 Ιανουαρίου στο Στρασβούργο, στις 21 Ιανουαρίου το πρωί στις Βρυξέλλες και 3 Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο. Όσον αφορά τη διερμηνία των συνεδριάσεων αυτών, να σας πω ότι δεν θα υπάρχουν δεν θα υπάρχει δανέζικη διερμηνία στις 16 και 17, φιλανδικά, στονικά, μαλτέζικα και κροατικά όμως επίσης δεν θα υπάρχουν. Σας ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση και τώρα περνάμε στην έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της 3ης Οκτωβρίου 2013 και 17ης Οκτωβρίου 2013. Εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσει μέχρι το τέλο τη αυριανή συνεδρίαση, θα θεωρήσω ότι τα πρακτικά έχουν εγκριθεί. Περνάμε τώρα στο σημείο 5 της ημερησίας διάταξης. Και εδώ θα ήθελα να καλωσορίσω την Αντιπρόεδρο Επίτροπο κυρία Ρέντινγκ για μια ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση σε θέματα ποινική δικαιοσύνη. και πληροφορίε για τη συνέχεια που δόθηκε στο Συμβούλιο Δικαιοσύνη και Εσωτερικών Υποθέσεων τη 5η και 6η Δεκεμβρίου 2013. Κυρία Ρέντινγκ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Με χαρά μου βρίσκομαι πάλι ανάμεσά σα. Την περασμένη εβδομάδα συμμετείχα στην ε, ακρόαση για τις αποκαλύψεις σχετικά με την NSA και συζητήθηκαν τα βήματα που χρειάστηκαν για την ενίσχυση της προστασίας προσωπικών δεδομένων των πολιτών μας, ιδιαίτερα όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο όμως αυτές. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τη μεταρρύθμιση της προστασίας δεδομένων στο εσωτερικό της Ένωσης. Εμείς, αυτό σημαίνει δηλαδή το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταφέραμε να θέσουμε θέματα στην ημερήσια διάταξη προστασίας δεδομένων και αυτό είναι ιδιαίτερη σημασία και για τους πολίτες μας και για τις επιχειρήσεις μας στην ε, ψηφιακή οικονομία. Έχουμε εργαστεί με όραμα και με αποφασιστικότητα και θα ήθελα εδώ να σας συγχαρώ για την ε, αποφασιστική ψηφοφορία σας τον Οκτώβριο. Έχουμε καταφέρει πολλά μαζί και είναι πολύ σημαντικό η ψηφοφορία στην Ολομέλεια να διεξαχθεί πολύ πριν την διακοπή για τις ευρωεκλογέ, έτσι ώστε να αναλογιστούμε και να σκεφτούμε αυτά που έχουν γίνει. Εδώ θα ήθελα να πω ότι λυπάμαι για το ότι δεν καταφέραμε να Έχουμε την ίδια αποφασιστικότητα στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης του Δεκεμβρίου. Όχι μόνο δεν προχωρήσαμε, αλλά πιστεύω πως ε, οπισθοχωρήσαμε. Και πιστεύω πως η μόνη έξοδος είναι στα χέρια της Ελληνικής Προεδρίας. Και η Ελληνική Προεδρία έχει θέσει την ε, μεταρρύθμιση της προστασίας δεδομένων ως ε, μία από τις κυριότερες προτεραιότητές της. Είμαι σίγουρη πως αυτό θα δώσει όφηση στο θέμα αυτό. Η Ελληνική Προεδρία θα ήθελε να εγκριθεί το νέο πακέτο το Μάρτιο και αυτό το στηρίζω απόλυτα. Ελπίζω λοιπόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει παρόμοια άποψη όσον αφορά τον Μάρτιο. Τώρα, θα ήθελα σήμερα να μιλήσω για έναν άλλο κοινό στόχο, κάτι το οποίο επεξεργαζόμαστε πολύ καιρό, τα δικονομικά δικαιώματα και τις κοινέ ασφαλιστικές δικλείδες για τους ύποπτους σε ποινικέ δίκες. Έχουν γίνει ακροάσεις και στην αρχή των ακροάσεων αυτών σας υποσχέθηκα να γίνει πρόοδος και έχει γίνει αρκετή πρόοδος. Έχουμε στα χέρια μας τρεις οδηγίες, το δικαίωμα σε διερμηνία και μετάφραση, το δικαίωμα στην πληροφόρηση όσον αφορά τις ποινικέ ε, διαδικασίες, δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο, έχουμε ενισχύσει τα δικαιώματα των θυμάτων και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας για την συνεχή σας στήριξη. Όχι μόνο, έχετε, όχι μόνο όσους έχετε συνεργαστεί για αυτό, αλλά όλους, διότι έχουμε τώρα κάποια ορόσημα στην προστασία των δικαιωμάτων. Επίσης θα, θα παρακολουθούμε πολύ στενά την εφαρμογή τους στην Εθνική Νομοθεσία. Την, στις 27 Νοεμβρίου κατέθεσα συμπληρωματικά δικονομικά δικαιώματα. Ένα τέτοιο πακέτο λοιπόν το οποίο αποτελείται από τρεις οδηγίες και δύο συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταρχάς, τεκμήριο αθωότητας. Αυτό ίσως σας ε, φαίνεται πολύ απλό, δεν είναι όμως δεδομένο σε καμία περίπτωση. Θα έπρεπε πάντα ο κατήγορος να πρέπει να αποδείξει την ενοχή και όχι ο ύποπτος να αποδείξει την αθωότητά του ένας ύποπτος δεν μπορεί να θεωρείται ένοχος εάν δεν του έχει δοθεί ποτέ η ευκαιρία να υπερασπιστεί τον εαυτό του σε μια δίκη. Και κανείς δεν θα πρέπει να υποθέτει ότι η σιωπή του κατηγορούμενου είναι και δήλωση ενοχής. Επίσης, έχουμε ασφαλιστικές ειδικλίδες όσον αφορά τα παιδιά που εμπλέκονται σε ποινικέ διαδικασίες, διότι όπως ξέρετε τα παιδιά πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν τις συνέπειες ε, των πράξεων τους και γι' αυτό δεν θα έπρεπε να υπάρχει δυνατότητα τα παιδιά να αρνούνται το δικαίωμα υπεράσπισης από δικηγόρο. Πάντα τα παιδιά θα πρέπει να έχουν έναν δικηγόρο δίπλα τους και επίσης να προστατεύονται και από άλλες διατάξεις όσον αφορά για παράδειγμα την πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματά τους, συνοδεία από γονείς οικειδαιμόνες, μαγνητοφώνηση των ε, ανακρίσεων και διάφορα άλλα μέτρα σχετικά με την υπεράσπιση την ελευθερία, της ελευθερίας. Προστασία για δίκη και δίκαιη δίκη και προστασία της κοινωνικής τους ένταξης. Μετά από, μέσα από τις ε, συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη να παράσχουν δικλείδες ασφαλείας και για, άλλους, ε, για άλλες κατηγορίες υπόπτων, για παράδειγμα άτομα με σωματική ή πνευματική αναπηρία. Τρίτον, έχουμε προτείνει μια οδηγία για προσωρινή νομική αρρωγή που θα καλύπτει τα αρχικά στάδια μιας ε, δίκης σε περιπτώσεις που οι ύποπτοι στερούνται βασικά δικαιώματα. Επίσης θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι κάθε ύποπτος έχει πρόσβαση σε νομική αρρωγή αφότου συλληφθεί και στην χώρα σύλληψης και στη χώρα εκτέλεσης ε, του εντάλματος. Και επίσης υπάρχουν κοινά κριτήρια τα οποία θα, θα αποφασίζουν εάν κάποιος έχει το δικαίωμα νομικής αρρωγής έτσι ώστε να προωθηθεί η σύγκληση των νομικών συστημάτων και να προωθηθεί και η εμπιστοσύνη. Ξέρω πως ε, είναι προχωρημένη ώρα, αλλά είμαι σίγουρη ότι η Επιτροπή σας θα εργαστεί για αυτό το πακέτο και ξέρω επίσης πως ε, βρισκόμαστε στο τέλος της θητείας, αλλά είμαι σίγουρη πως θα εργαστείτε για να δώσετε στην επόμενη Επιτροπή ένα καλό αποτέλεσμα. Τώρα όσον αφορά την οδηγία για την πλαστογραφία και, τα... και την παραποίηση. Ελπίζω το Κοινοβούλιο να ορίσει τη θέση του σύντομα, έτσι ώστε οι δύο οδηγίες να εγκριθούν πριν από το καλοκαίρι του 2014. Αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για τον έξω κόσμο, ότι το Κοινοβούλιο δηλαδή εργάζεται για την προστασία των πολιτών, των αγαθών και της αγοράς της Ευρώπης. Επίσης ελπίζω η δουλειά σας να ανταποκριθεί στις προσδοκίες και στην, στη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την καταπολέμηση των νέων μορφών εγκλήματος, διότι διαφορετικά θα συνεχίσουν να καταλήγουν τα χρήματα των φορολογούμενων σε λάθος τσέπες. Τέλος τώρα θα ήθελα να καλωσορίσω την πρόθεση των κύριων Ποστάσιεβιτς και Μπεσερίλ να εγκρίνουν σε πρώτη ανάγνωση την, ε, το πακέτο για τις ε, ναρκωτικές ουσίες. Τέλος, όσον αφορά τον πίνακα επιδόσεων ε, σε θέματα δικαιοσύνης. Να σας ενημερώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει αυτό το εργαλείο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ο πίνακας επιδόσεων θα παρέχει αξιόπιστα δεδομένα όσον αφορά την ποιότητα και την ε, ανεξαρτησία και αμεροληψία των εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης, αντιμετωπίζει εξίσου όλα τα κράτη-μέλη και θα παρέχει μια συνολική εικόνα της λειτουργίας των νομικών και δικαστικών συστημάτων. Το πίνακας αυτός επιδόσεων είναι ένα εργαλείο, δεν είναι ούτε νομικό μέσο, ούτε τίποτα διαφορετικό, ούτε προς καλοπισμό. Είναι ένα εργαλείο που θα μας βοηθήσει, θα βοηθήσει και το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις εργασίες του. Πέρυσι συζητήθηκε η πρόσβαση στα δεδομένα. Φέτο, κατόπιν αίτηση τριών κρατών μελών, που είναι επίση μέλη του Συμβουλίου τη Ευρώπη, τη Ισπανία, του Ηνωμένου Βασιλείου και τη Σουηδία, το ΣΕΠΕΣ δεν εγκρίθηκε. δυστυχώ. τα κράτη-μέλη αυτά χρησιμοποίησαν μια απόφαση για να μπλοκάρουν προσωρινά την απόφαση και να θέσουν υπό αμφισβήτηση των πίνακα επιδόσεων της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Αν και μια μεγάλη μερίδα των κρατών μελών στηρίζει τον πίνακα αυτόν. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη στον δικαστικό τομέα για να παρακάμψουμε το με αυτό και να υπογραφεί η σύμβαση. Το επιτελείο μου αύριο θα συνεδριάσει για αυτά τα σημεία, με, τα σημεία επαφή των κρατών μελών, έτσι ώστε να συζητηθεί ο πίνακα επιδόσεων για το 2014. Τώρα, στην Επιτροπή αυτή, όλα αυτά τα χρόνια, εσείς είστε η κινητήριος δύναμη που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και την ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών. Γνωρίζετε ότι κάποια κράτη-μέλη προσπαθούν να αμφισβητήσουν αυτό το θεμελιώδες δικαίωμα, αυτή τη θεμελιώδη ελευθερία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ξεκάθαρη όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο να σας πω και ότι αμφισβητείται έντονα και από τους πολίτες των κρατών μελών στις ε, δημοσκοπήσεις ε, που έχουμε κάνει, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν την ελευθερία της ε, μετακίνησης ένα από τα ύψιστα και πιο σημαντικά δικαιώματα που έχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, οι αντιλήψεις της κοινή γνώμης δεν είναι βασισμένες σε γεγονότα. Και εμείς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ε, αντιλήψεις και τις ανησυχίες των κρατών μελών και των κυβερνήσεων, διότι ξέρουμε πως όντως υπάρχουν περιπτώσεις καταχρήσεων. Γι' αυτό ε, υπήρξε μια σύσταση της ε, Κομισιόν για την ελευθερία της μετακίνησης η οποία περιλαμβάνει διατάξεις που επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να καταπολεμήσουν περιπτώσεις κατάχρησης και απάτης στην ελεύθερη μετακίνηση. Επίσης έχουμε προτείνει στα κράτη-μέλη να, τους, να τα βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά με ένα σχέδιο δράσης πέντε σημείων. Συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη για την δημιουργία ενός εγχειριδίου όσον αφορά τους ε, συμβατικούς γάμους αυτό είναι ένα φαινόμενο που έχουν ε, να αντιμετωπίσουν πάρα πολύ συχνά οι δημόσιες υπηρεσίες. Ταυτόχρονα συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη για να δημιουργηθεί ένας οδηγός σχετικά με την συνήθη διαμονή, η οποία πολλές φορές ε, εμπλέκεται σε περιπτώσεις καταχρήσεων συστηματών κοινωνικής ασφάλισης. Συζητήθηκε επίση το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και η χρήση του για την επόμενη περίοδο. Προωθήθηκε η συνεργασία ανάμεσα σε εθνικέ και τοπικέ αρχέ και το 2014 στι 11 Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί ένα μεγάλο συνέδριο για Δημάρχου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τους εξηγήσουμε και να τους αναφέρουμε τι δυνατότητες έχουν όχι μόνο νομικά αλλά και ως προς τη χρήση των κοινωνικών ταμείων. Επίσης, Έχουμε διάφορα προγράμματα κατάρτισης για την προώθηση της ελεύθερης μετακίνησης, προγράμματα που απευθύνονται στις τοπικές αρχές. Έχουμε μεγάλη στήριξη από το Συμβούλιο, μεγάλη πλειοψηφία υπουργών εσωτερικών μας υποστηρίζουν και αυτό ε, φάνηκε στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Και τώρα θα αρχίσουμε σιγά σιγά να εφαρμόζουμε το ε, σχέδιο δράσης πέντε σημείων. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία στο Κοινοβούλιο να το συζητήσουμε δημόσια και ε, είναι στα χέρια σας να αλλάξετε την άποψη της εκείνης γνώμη και να υπερασπιστείτε ένα από τα πιο σημαντικά δικαιώματα που έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Επίσης, θα ήθελα να σας ενημερώσω για ένα σημαντικό επίτευγμα όσον αφορά την κοινωνική συμπερίληψη των Ρωμά. Ίσως φαίνεται απίστευτο, αλλά το Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την ε, σύσταση του Συμβουλίου στις 9 Δεκεμβρίου και πιστεύω πως αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το επίτευγμα σημαίνει ότι χρειάζεται πλέον συντονισμένη δράση και αυτό έχει αναγνωριστεί από τα κράτη-μέλη. Και αυτό δεν είναι μόνο επιτυχία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που κατέθεσε την πρόταση, είναι και μια επιτυχία του Κοινοβουλίου, το οποίο ανέκαθεν στήριζε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στην ε, συμπερίληψη των Ρωμά και δίνει μια ελπίδα πλέον στους Ρωμά. Και ελπίζω να έχω την ε, στήριξή σας και την έγκρισή σας πολύ σύντομα. Τώρα, Για το μέλλον. Το Μάρτιο η Κομισιόν θα ήθελε να δημοσιεύσει μία σύσταση για την δικαστική συνεργασία. Θέλουμε να αποφύγουμε την άγρα δικαστηρίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται μία όρημη ευρωπαϊκή πολιτική και δεν υπάρχει λόγος να μας καθυστερήσουν τα οποιαδήποτε χρονοβόρα προγράμματα, όπως το πενταετές πρόγραμμα. Είμαστε πλέον χρόνια μετά την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας και πρέπει πραγματικά να χρησιμοποιήσουμε, να εκμεταλλευτούμε τα πλέον εκτήματα που μας δίνει αυτή. Γι' αυτό λοιπόν ελπίζω το σχέδιο έκθεσης για την ενδιάμεση αναθεώρηση του προγράμματος της Χόλμης να ανακλά αυτήν την βούληση. Επίσης, έχουμε μία ολοκληρωμένη προσέγγιση που ε, συμπεριλαμβάνει όλους τους, ε, τους ε, συμμετέχοντες, όλους τους φορείς. Σε ένα σχετικό συνέδριο, να σας πω ότι είχαμε πάνω από 600 συνέδρους και εδώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την στήριξή σας. Τέλος, θα ήθελα να πω δύο λόγια για το κράτος δικαίου. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Μπαρόζο στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται μια ανακοίνωση που θα παρουσιαστεί την άνοιξη του 2014. Προετοιμάστηκε ένα έγγραφο για το πλαίσιο του κράτους δικαίου, έτσι ώστε να αρχίσει η συνεδρίαση, η συζήτηση, με συγχωρείτε, και ελπίζω να συζητηθεί το θέμα στα πλαίσια της έκθεσης Μισελ για τα, ανθρω... για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτά προς το παρόν. Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, ελπίζω να συνεχίσουμε την καλή, εξαιρετική καρποφόρο συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Mm, Uh, Ευχαριστώ κυρία Αντιπρόεδρε. Τώρα έχουν ζητήσει το λόγο κάποιοι συνάδελφοι. Πρώτα οι συντονιστές, η κυρία Αργεντινή, ο κύριος Κιρκόπφ. μετά ο εισηγητής για την προστασία δεδομένων ο κύριος Άλμπρεκτ και τα μέλη που έχουν ζητήσει η κυρία Σίγμπελ, η κυρία Λότφορντ, Ντελόγκ, Γκούντ, Hintveld και Μπράουν. Ναι, ναι, μα είπα το όνομά σας ήδη. Αυτός είναι ο κατάλογος των αγορητών. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στους αδέλφους για δύο λεπτά για να μείνουμε εντός του χρονικού πλαισίου. Κύριε Αργεντίνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. θα ήθελα να μιλήσω για την ε, νομική αρρωγή. Είμαστε ικανοποιημένοι για την προσέγγιση, αλλά θέλω να ακούσουμε την άποψή σα ε, σχετικά με τα όσα συμβαίνουν στη χώρα μου, την Ολλανδία, όπου οι δικηγόροι αυτή τη στιγμή ε, διαμαρτύρονται κατά και θεωρούν ότι οι δικαστές έχουν δυσκολίες να αντιμετωπίσουν τον όλο όγκο των εργασιών για τις, που προκύπτουν μετά από τις διάφορες περικοπές και ε, υπουργό Δικαιοσύνης προτείνει ένας κατηγορούμενος ο οποίος περνάει όχι, θα αρχίσω να μιλάω Ολλανδικά γιατί είναι πολύ νομική φύση το ζήτημα. Θα... Ένας ύποπτος λοιπόν, ο οποίο έχει δικαίωμα σε μια... στο δικαίωμα τη προσφυγή, μπορεί να ζητήσει, μάλλον η δικαιοσύνη μπορεί να τον στείλει στη φυλακή, ενώ η έφεσή του δεν έχει ακόμα εξεταστεί. Φυσικά λυπάμαι για κάτι τέτοιο, μέχρι τώρα η χώρα μου ήταν ένα παράδειγμα, ένα υπόδειγμα μάλλον σε θέματα δικαιοσύνη και διερωτώ με εάν υπό το φως των προτάσεων που κάνατε κυρία Αντιπρόεδρε για τη βελτίωση της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά σε ό,τι τα δικαιώματα των υπόπτων, τι πιστεύετε για την εξέλιξη στις κατοχώρες. Κύριε Κύρκοφ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την ε, κυρία Επίτροπο. Να ξεκινήσω λέγοντας ε, ότι κάποιες παρατηρήσεις της Επιτρόπου με ενθάρρυνε για να αντιμετωπίσουμε κάποιες ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, που μας πλήττουν μάλλον, σε ό,τι φορά τώρα τους Ρώμα, να πω πρώτον Πιστεύει η Επίτροπος ότι πρόσφατες δηλώσεις σχετικά με την κυβέρνηση της Ηνωμένου Βασιλείου και παραθέτω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο καταστρέφει την ελεύθερη διακίνηση. Νομίζουμε ότι αυτά είναι λόγια τα οποία μπορούν να τύχουν τη στήριξη του, του Βρετανικού λαού προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεύτερον πολύ συζητημένο θέμα είναι το ζήτημα των, των διαφόρων φακέλων που φορούν στους, στην καταπολέμηση της ε, παραποίησης του ευρώ και τις σχετικές κυρώσεις. Μπορούσε η Επίτροπος να μας ε, αναφέρει σχετικά με την αρμόνιση αυτών των ποινών και τι πρόοδο είδαν να πετυχαίνεται στα κράτη-μέλη τα οποία επιθυμούσαν να αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτά τα ζητήματα. Κ. Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσω για την πληρέστατη παρουσίαση των γεγονότων και σε ό,τι φορά τα ελάχιστα στάνταρ να πω ότι πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση είναι ένα πολύ καλό βήμα αυτό της πρότασης των νέων μέτρων θα ήθελα να προχωρήσουμε ταχύτατα διότι υιοθετήσαμε και το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Ερεύνης και φυσικά απαιτούνται κάποια ελάχιστα στάνταρ στον τομέα της ποινική δικαιοσύνης. ό,τι φορά τώρα την προστασία δεδομένων θα ήθελα να εκφράσω την απογοήτευσή μου και νομίζω ότι μπορώ να το κάνω εξ ονόματος όλων των συναδέλφων, διότι το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να συμφωνήσει για την σχετική μεταρρύθμιση και έτσι ο κανονισμός και η οδηγία για την προστασία δεδομένων παραμένουν ως έχουν και εμείς είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις το συντομότερο ως Κοινοβούλιο. Θέλουμε να το χωρίσουμε τάχιστα και πιστεύω πως το Συμβούλιο όπως το θέμα του non-stop shop, one-stop shop, θα έπρεπε να πάρει κάποιες αποφάσεις. Το ψηφίσαμε ομόφωνα, αυτό κάτι το οποίο βελτιώνει το σύστημα και νομίζω θα πρέπει να το λάβει υπόψη του αυτό το Συμβούλιο. Όπως σας είπε, είμαι κάπως απογοητευμένος που αυτό δεν συνέβη και είμαι έτοιμος να εξηγήσω καλύτερα την θέση μας προς το Συμβούλιο προκειμένου να πετύχουμε συνένεση το συντομότερο τώρα για το ζήτημα του ορισμού του Ευρωπαίου Επόπτη Δεδομένων και εδώ με ανησυχεί το ζήτημα γιατί ακούω διάφορες φήμες Κανονικά θα πρέπει να είμαστε τώρα σε θέση να ενημερωθούμε αναφορικά με τον διορισμό αυτών και σχετικά με τη shortlist Γνωρίζω ότι είναι αρμοδιότητα την Επιτρόπου Σεύκοβιτς, ε, Επιτρόπου αλλά θα ήθελα να δώσει προφορίες το συντομότερο προς το Κοινοβούλιο αναφορικά με τον εν λόγω διορισμό. Ευχαριστώ κύριε Άλμπρεχτ, κυρία Σίμπελ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να τοποθετηθώ και τα ακόλουθα. Καταρχάς, τα οικονομικά δικαιώματα. Να πω ότι Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις περαιτέρω προτάσεις που έχει κάνει, όμως θα ήθελα να συμπληρώσω και εγώ την κυρία Σαρτζεντίνη λέγοντας ότι χρειάζεται μια στενή συνεργασία αστυνομία και ε, δικαστικού σώματος και τα κονδύλια και τα μέσα που έχουμε στην ε, διάθεση μας δεν επαρκούν. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να βελτιώσουμε τα δικονομικά δικαιώματα και τα δικαιώματα των κατηγορουμένων. Γι' αυτό δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται τα κράτη-μέλη να κάνουν λόγο για περικοπές στο θέμα αυτό. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω και ελπίζω οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μας πάνε λίγο παραπέρα. Τώρα, όσον αφορά την ελεύθερη μετακίνηση. Η ελεύθερη μετακίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι όντως ένα από τα βασικότερα δικαιώματα που έχουμε, θεμελιώδης αξία. Και αυτά που έχω ακούσει προς το παρόν από το Ηνωμένο Βασίλειο και από την Γερμανία είναι απαράδεκτα κατά την άποψή μου. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με την ελεύθερη μετακίνηση, δεν έχουμε μόνο μάλλον προβλήματα, δεν έχουμε προβλήματα με την μετακίνηση των ε, Ρωμά. Υπάρχουν συγκεκριμένα όμως ε, μέρη, συγκεκριμένε γειτονιές σε πόλεις οι οποίες ε, γειτονιές αυτές έχουν προβλήματα, υπάρχει μεγάλη προσέλευση Ρωμά και αυτές οι περιοχές θέλουν οικονομική στήριξη και αυτό δεν μπορεί μόνο να το αντιμετωπίσει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί και από τα κράτη-μέλη τα ίδια, γιατί είναι θέμα βασικών θεμελιωδών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, το τρίτο σημείο είναι το εξή, κυρία Ρέντινγκ, αναφερθήκατε στην προστασία δεδομένων και το σκάνδαλο με την NSA. Και εδώ θα ήθελα να συμφωνήσω με τον συναδέλφο κύριο Άλμπρεχτ. Υπάρχουν φήμες ε, οι οποίες οργιάζουν και τώρα πραγματικά βρισκόμαστε σε... Βρισκόμαστε σε αδέξοδο από τις 43 προτάσεις που έχουν γίνει για υπεύθυνο για το θέμα αυτό. Έχουμε καταλήξει σε 5. Καταρχάς, έχει προταθεί ο υποψήφιος που θα αναλάβει το θέμα αυτό να είναι κάποιος φιλικά προσκύμενος προς τις Ηνωμένε Πολιτείε. Δεν ξέρω αν είναι φήμη αυτό ή αν είναι πραγματικότητα, όμως θα ήθελα να μας ενημερώσετε ε, λεπτομέρως σχετικά. Έπειτα, υπάρχουν τρία ονόματα καθώς ακούω που έχουν προταθεί και εγώ πιστεύω πως δεν αρκούν τρία, τρεις μόνο υποψήφοι από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν αρκούν μόνο τρεις. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Ρέντινγκ να μου επιβεβαιώσει ή να μου αρνηθεί τι εφήμε. Κυρία Λάντφορντ. Ευχαριστώ. Να σας ρωτήσω σχετικά με την προνόμη δικαιοδοσία για τα δικονομικά δικαιώματα. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά κρατημέλη και μεταξύ αυτών το ΙΤΑΒ που σε κάποιες ε, περιπτώσεις ε, δεν διαφωνούμε και από ό,τι καταλαβαίνω το δικαστήριο του Στρασβούρου στην υπόθεση Κόνραντ αναγνώρισε πως ε, το νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου πετυχαίνει τη σωστή ισορροπία. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε μια κατάσταση όπου η επεξήγηση απαιτείται, τότε η σιωπή θα έχει την σημασία της όταν θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το δικαστήριο. Λοιπόν, κανένα άποψή μου είναι ε, το, η απόφαση του δικαστήριου του Στρασβούργου δεν επιτρέπει σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις να γίνει κάτι τέτοιο. Η Κομισιόν υπέβαλε την πρότασή της, ότι δηλαδή δεν μπορεί να ε, συναχθούν κάποια συμπεράσματα ένεκα της σιωπής του κατηγορημένου ή πιστεύει πως δεν θα πρέπει να λαμβάνει η απόφαση του ασβούλου υπόψη, διότι θεωρώ ότι υπάρχουν περιπτώσεις ε, κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται. Εγώ συνεργάζομαι με τους ε, σκιώδες ηγητές ε, πάνω στο ζήτημα του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Μία από τις ιδέες που προτείνουμε είναι και θα ρωτήσουμε την Κομισιόν να κάνει μια πρόταση νομοθετικού περιεχομένου για οριζόντια μέτρα ώστε να καλυφθούν μέτρα για όλα τα μέσα αμοιβές αναγνώρισης όπως το θέμα της αναλογικότητας που έχουμε στην Ευρωπαϊκό Ένταλμα Έρευνας και διάφορες άλλα νομικά μέτρα μπορούν αυτά να εξεταστούν πριν να εφαρμοστεί το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Έχει η Κομισιόν μια άποψη αναφορικά με οριζόντια μέτρα, αναφορικά με την αμοιβαία αναγνώριση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με την κυρία, Αργεντίνη σε θέματα νομικής, δικαστικής αρρωγής και ε, τα σχετικά δικαιώματα. Ελπίζω πως η Επίτροπος Ρέντινγκ να ενεργήσει επί του θέματος, διότι όντως το ζήτημα είναι κατεπήγον. Ε, δεύτερον, έμαθα από τα μέσα ενημέρωσης πως η Ρουμανία υιοθέτησε μια νομοθεσία η οποία αντιβαίνει σε όλα αυτά. και νομίζω ότι αυτό δημιουργεί μια κατακραυγή από πλευρά ρουμανικού λαού. Ποιε είναι όμω οι συνέπειε ε, όλων αυτών κατά τη ε, ελεύθερη διακίνηση, ελεύθερη κυκλοφορία. Ποια είναι τα μέτρα λοιπόν που ο Επίτροπο Ρέντινγκ προτίθεται να λάβει, διότι νομίζω ότι το ζήτημα έχει ιδιαίτερη σημασία. Κάτι ακόμα. Ο Ευρωπαίος εισαγγελέα ε, Φυσικά έχουμε την ανακοίνωση της Επιτροπής Περί αυτού αλλά θα ήθελα να γνωρίζω τι αξιολόγηση κάνει ε, η κυρία Ρέντινγκ για τη στάση του Συμβουλίου. Πώς ε, πιστεύει να ε, εφαρμοστεί η ενισχυμένη συνεργασία και ποιο θα είναι τα συμπεράσματα, τα αποτελέσματα μιας ενισχυμένης συνεργασίας για την Όλαφ. Και αυτό που είπε ένας συνάδελφος σχετικά με τις ελάχιστες κυρώσεις, Νομίζω ότι υπάρχει ευρύτατη συνένεση στο Κοινοβούλιο. Δηλαδή όλοι διαπιστώσαμε πως προτάσεις της ε, Κομισιόν δεν είχε ακόμα οριμάσει και θα ήταν σκόπιμο επί του θέματος η Κομισιόν να μας στείλει ένα νέο έγγραφο εργασίας, ίσως κάτι το οποίο θα προέρθει από τους υπαλλήλους μεν, αλλά πώς η Κομισιόν κατέληξε σε αυτήν την απόφαση ότι χρειάζονται ελάχιστες ποινές ανεξάρτητα από, το, τη σημασία, τη σοβαρότητα του εγκλήματος που διπράκτων. Πολλά υπόθηκαν. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Δύο συμπληρωματικές ερωτήσεις. άποψή μου, η δικαστική δικαιοσύνη είναι απαραίτητο να τη χάνει αμοιβές αναγνώρισης ε, στο πλαίσιο της συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να επεκτείνεται τα δικαιώματα της Fundamental Rights Agency στα κράτη-μέλη. Η άλλη ερώτησή μου σχετίζεται με την ανακοίνωση σχετικά με το κράτος δικαίου είπατε ότι προτίθεστε τον Απρίλιο, μάλλον την Άνοιξη να καταλήξετε σε κάτι τέτοιο. Το Κοινοβούλιο επανειλημμένα έχει ζητήσει κάτι τέτοιο. Θα ήθελα να γνωρίζω μια ακριβέστερη ημερομηνία ή δυνατόν για την λόγω ανακοίνωση του θέμα είναι σημαντικό διότι θα ήθελα να γνωρίζω αν κατά πόσον το Κοινοβούλιο με, σε αυτή τη θητεία θα μπορέσει να την εξετάσει. Αν συμβεί αρχές Μαρτίου θα είναι δυνατόν. Αν φτάσει αργότερα τότε θα είναι κατά το μάλλον ή τον αδύνατον. Θα ήθελα να γνωρίζω λοιπόν μια πιο ακριβέστερη ημερομηνία. Ευχαριστώ. Um, the Commissioner mentioned... Η Επίτροπος ε, μίλησε για δικονομικές αλλαγές σε σχέση με τη νομική αρρωγή στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, αλλά δεν λάβαμε υπόψη στη περίπτωση αυτή τα αποδεικτικά στοιχεία και την εξέτασή τους ζητώντας, προβάλλοντας αυτό το ένταλμα ε, με βάση ανεπαρκή στοιχεία, διότι στη δική μου χώρα τα δικαστήρα μπορούσαν να απορρίψουν το αίτημα εάν δεν υπήρχαν, δεν υπήρχαν επαρκείς αποδείξεις όπως στην περίπτωση ε, μιας ποινική δίκης. Μιλήσατε για την ελεύθερη διακίνηση και είπατε ότι είναι το πιο ε, αξιόλογο ε, δικαίωμα σε αυτή την περίπτωση. Τη στιγμή που μιλάμε για συγκρίσιμο ε, πλούτο, δεν ξέρω κατά πόσο η κλίμακα είναι ίδια. Όταν αυτά τα δικαιώματα αφορούν χώρες με διαφορετικό ΑΕΠ, επί τρία ή περισσότερο, τότε θα υπάρχει ε, μεγάλος φόρτος, ιδιαίτερα ως προς τις κοινωνικές παροχές και αυτό αφορά ιδιαίτερα το εργατικό δυναμικό ορισμένων χωρών λόγω μετανάστευσης. Είναι πολύ δύσκολο να σκεφτούμε ότι οι πολίτες θεωρούν ότι η ελεύθερη διακίνηση είναι τόσο ή περισσότερο σημαντική ε, σε σχέση με άλλα βασικά δικαιώματα όπως το δικαίωμα ε, έκφρασης, ελεύθερης έκφρασης ή του συνεταιρίζεστε. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν ίσα δικαιώματα σε όλα τα κράτη-μέλη. Ιντφελτ. Ευχαριστώ. Έχω μόνο μερικές ερωτήσεις. Δέχομαι το, τα πενταετή προγράμματα που προβάλλατε και δέχομαι τις ανησυχίες που εκφράστηκαν σε σχέση με τον διορισμό του το επόπτη προστασίας προσωπικών δεδομένων. Το δεύτερο ερώτημα αφορά το αίτημα του Κοινοβουλίου με βάση την έκθεση Λούνατσεκ, το αίτημα ενός οδικού χάρτη για τα δικαιώματα των ΛΟΑΔ. Νομίζω ότι θα πρέπει να προκριθεί μια πρόταση το σύντομότερο δυνατόν και να μην τα αφήσουμε στις δικαστικές αρχές γιατί υπήρχαν ε, συγκεκριμένες επικής, όχι αλλά σωστές και ευνοϊκές αποφάσεις για τα δικαιώματα των ΛΟΑΔ. Αλλά δεν μπορούμε να παίρνουμε πολιτικές αποφάσεις εμείς οι ίδιοι. Και ένα τελευταίο το οποίο θα συζητήσουμε αργότερα είναι η διαφάνεια και η πρόσβαση στα έγγραφα. Δεν είναι το δικό σας χαρτοφυλάκιο βεβαίως, αλλά είναι κοινή ευθύνη να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει πραγματική διαφάνεια και αυτό είναι ζωτική σημασίας και για τη δική σας πολιτική διότι είναι αναπόσπαστο τμήμα των ε, βασικών ελέγχων που διενεργούνται και σε περίπτωση στασιμότητας τι προτείνεται έτσι ώστε να επανακινηθεί η διαδικασία. Μπάουερ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να υποβάλω ε, μια ερώτηση σαν αυτή που προηγήθηκε. Επειδή στην καθημερινή ζωή αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις και επειδή θέλουμε να εξευρεθούν λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η κατάσταση των ανηλίκων, των παιδιών είναι ύψης της σημασίας. Ξέρουμε ότι γίνονται μεικτοί γάμοι, αλλά έχουμε να αντιμετωπίσουμε και σωρία διαζυγίων. Τα παιδιά αυτά λοιπόν είναι σε μια ιδιαίτερα ευάλωτη θέση τις περισσότερες φορές. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έθεσε το ερώτημα του κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιληφθεί αυτού του ζητήματος και κατά πόσο το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προβεί σε συστάσεις για το δικαίωμα επίσκεψης και ούτω καθεξής. Πρόκειται για καθημερινά ζητήματα τα οποία πρέπει να διευθετηθούν. Δηλαδή προσχωρούμε σε αυτές τις συμβάσεις, αλλά πολλές φορές δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν την τη συνθήκη της Λισαβόνας. Άρα το ερώτημα είναι κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να προωθήσει και αυτή την ε, πτυχή του ζητήματος. Ο κύριος Φως. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σχετικά με Στη συνέχεια και το μέλλον του Ευρωπαίου Πόπτη Προστασίας Δεδομένων. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε κάποιες λεπτομέρειες γι' αυτό. Έπειτα, ε, τι θα γίνει με την ε, περαιτέρω εξέλιξη του φακέλου για την προστασία των δεδομένων πώς σκέφτεται η Κομισιόν, πώς σκέφτεται το Συμβούλιο να προχωρήσει. Μας είπατε ότι τα πράγματα δεν φαίνονται και τόσο καλά και ότι έχουν παρατηρηθεί οπισθοχωρήσεις αντί για πρόοδος. Τι έχετε λοιπόν να πείτε γι' αυτό και τρίτον όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Eurojust και το μέλλον τους. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω με βάση τις εξελίξεις στο Συμβούλιο ότι ποιο είναι το μέλλον της ε, Eurojust προβλέπετε κάποια συνεργασία, υπάρχει θέληση για συνεργασία, υπάρχουν ιδέες ή προτάσεις για το πώς θα βελτιωθεί η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και πώς θα συμπεριληφθούν και τα κράτη-μέλη περισσότερο στα αυτήν. Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις από τα μέλη. Δίνω το λόγο σε εσάς. Ε, κυρία Αντιπρόεδρε, έχετε σωρία ερωτήσεων. Ναι, πράγματι, αλλά για μία φορά έχουμε λίγο χρόνο και έτσι μπορώ πραγματικά να απαντήσω όσο πιο διεξοδικά γίνεται. Σε σχέση με την νομική αρρωγή, στις προτάσεις που έχω υποβάλει Προσπαθώ να προβάλλω εξειδικευμένες λύσεις, χωρίς όμως να μπω στις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών. Γι' αυτό εστίασα την ε, προσοχή μου στο γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει νομική αρρωγή έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να εξευρεθεί μια συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου σε έναν ε, ιδεατό κόσμο θα έπρεπε να επικρατήσει ομοφωνία κατά της ε, πρότασης. Θα ήθελα λοιπόν αυτοί που χρήζουν αρρωγής ή κρατούμενοι και στις απαρχές της ε, διαδικασίας να μπορέσουν να τύχουν αρρωγής. Και αυτό αφορά και το Ευρωπαϊκό Ένταλμα ε, σύλληψης. Αυτές οι προτάσεις ε, βρίσκονται επί τάπητος. Ε, κύριε Κίρκοπ, το, το ευεργέτημα αυτό που προβάλλατε, το έχουν, έχουν υποβάλει αυτή την ερώτηση και άλλα κράτη-μέλη. Για να είμαστε σαφείς, εμείς με βάση τα στοιχεία που μας έδωσαν τα κράτη-μέλη, προβήκαμε ε, σε μία ανάλυση, δηλαδή εάν υπάρχει θέμα ε, τέτοιου ευεργετήματος, ε, ποια είναι τα εμπλεκόμενα ποσά. Εσείς έχετε την έκθεση και έχετε τις λεπτομέρειες στην έκθεση που εξέδωσα. Βλέπετε ότι τα ευεργετήματα αυτά κατανέμονται στα κράτη-μέλη, ας πούμε ένα 85-90% στους, ε, σε αυτούς που κατέχουν την υπηκότητα, στους υπηκόους των κρατών μελών. Μεταξύ 0,4% και 1 ή 2% μιλάμε για το ευεργέτημα που προβάλλεται για Ευρωπαίους πολίτες. Και αυτό γιατί. Γιατί όσοι διακινούνται ελεύθερα, όσοι Ευρωπαίοι ε, διακινούνται ελεύθερα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το δικαίωμα για να εργαστούν. Ενώ σε ορισμένα κράτη-μέλη, και αυτό έχει ίσως σχέση με τρίτες χώρες, με υπηκόους τρίτων χωρών, τα ποσά που διατίθενται για τις ε, τρίτες χώρες ε, είναι κατά ε, επί 10 μάλλον πολλαπλάσια σε σχέση με αυτά που διατίθενται στους Ευρωπαίους πολίτες. Άρα ίσως ανακύπτουν προβλήματα στα κράτη-μέλη με βάση το εθνικό δίκαιο, διότι ορισμένοι εθνικοί νόμοι επιτρέπουν σε εκείνους που προσέρχονται σε ένα κράτος, άλλο κράτος μέλος, όχι στο κράτος προέλευσης, να ευεργετούνται από την πρώτη μέρα. Αυτό δεν εγγράφεται στην οδηγία. Η οδηγία αναφέρει ότι οι πίκοοι που θέλουν να παραμείνουν θα πρέπει να δείξουν ότι έχουν επαρκή εισοδήματα για να διαμείνουν. Τα μεγαλύτερα προβλήματα ανακύπτουν από ιδιαίτερα ευεργετικού νόμους στα κράτη-μέλη που δεν είναι ευρωπαϊκή Υφή, διότι το, τα κοινωνικά ευεργετήματα αφορούν το εθνικό δίκαιο. Γι' αυτό ζήτησα από τα κράτη-μέλη να δουν σοβαρά τι δεν κινείται σωστά στα κράτη-μέλη και να επανέλθουν, να προσγειωθούν δηλαδή κάπως και να δουν πού ακριβώς ανακύπτουν τα προβλήματα. Στην Υπουργική Συνάντηση των Υπουργών Εσωτερικών διαπίστωσα ότι μόνο ένα κράτος μέλος ζήτησε την αλλαγή της οδηγίας για την ελεύθερη διακίνηση. Τα άλλα κράτη-μέλη ζήτησαν βοήθεια αν υπάρχουν καταχρήσεις και αυτό ακριβώς έκανε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις προτάσεις που θέτει επιτάπητος. Ως προς τις ποινικέ ευθύνες και κυρώσεις, θυμάμαι, όταν μελετούσα πριν από την ακροασή μου και είδα τι είχαμε επιτάπητος τότε, ως προς το ποινικό σκέλος, το ποινικό δίκαιο, είχαμε να κάνουμε με κατασταλτικά μέτρα αποκλειστικά και αυτό είναι κατανοητό, διότι όλα είχαν γίνει χωρίς την αρρωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί μιλούσαμε για ε, εποχή πριν από τη συνθήκη της Λισαβόνας, από τους υπουργούς και μόνο μετά την 19η ε, Πρόκειται για μέσα και μηχανισμούς που ευτυχώς δεν εφαρμόστηκαν διότι δεν είχαν συνταχθεί σωστά, δεν υπήρχε μελέτη αντικτύπου, δεν είχε συνεργαστεί το Κοινοβούλιο και γι' αυτό δεν μπορούσαν να τύχουν εφαρμογής. Γι' αυτό ε, κατέστη αναγκαίο κάποια στιγμή να ανακύψει ένα άλλο στοιχείο που είναι τα δικαιοδοτικά δικαιώματα σε, ε, στα ποινικά καθαρά. Δηλαδή, πέρα από, τα, την καταστολή θα πρέπει να ε, προασπίσουμε και τα δικαιώματα του υπόδικου πριν ε, δικαστεί και μιλήσαμε για αμοιβαία αναγνώριση και εμπιστοσύνη. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη νομική βάση, την αναλογικότητα και την αρχή της επικουρικότητας. Και ακριβώς αυτό αποτελεί την κινητήριο δύναμη όλων των προτάσεων που, υπάρχουν, που έχει προβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με βάση τη διαθέσιμη νομική βάση, ο κύριος Άλμπρεχτ μίλησε για το ένταλμα έρευνας. Αυτό είναι ένα ζήτημα όπου έπρεπε να φτάσουμε σε μία εξισορρόπηση με τα δικαιοδοτικά δικαιώματα. Εγώ δεν προέβαλα αυτό το ένταλμα έρευνας. Ήταν μία ιδέα προ συνθήκης της Λισαβόνας. Καταλαβαίνετε τι δεν πάει καλά. Δεν με καλύπτει το κείμενο επιτάπητος και δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό το κείμενο ε, προωθήθηκε. Ε, ως προς τη μονοθυριδική προστασία δεδομένων, όλα συζητήθηκαν από πάνω προς τα κάτω, δεξιά, αριστερά τρεις φορές. Αυτό σημαίνει ότι το Συμβούλιο είναι έτοιμο να λάβει αποφάσεις, τα πράγματα όμως έχουν δυσχερανθεί. Και έχετε δίκιο, θα μπορούσαμε να ανατρέξουμε στην εργασία του Συμβουλίου επί Ιρλανδικής Προεδρίας και μετά να δούμε τι αποφάσισε το Κοινοβούλιο και να δούμε κατά πόσο υπάρχει συμφωνία Συμβουλίου ε, Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι είναι ευκταίο γιατί δεν χρειάζεται ε, να γίνουν νέες συζητήσεις. Όλα έχουν συζητηθεί ως προς την προστασία δεδομένων. Απλώς χρειαζόμαστε αποφάσεις, αν συμφωνούμε ή όχι. Με την καλή θέληση, με λίγη καλή θέληση, η ελληνική προεδρία θα προωθεί στο θέμα, διότι έχει ως προτεραιότητα, μία από τις προτεραιότητες της είναι και η προστασία δεδομένων. Άρα είναι κάτι το ε, ευκταίο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσει να βοηθήσει το Συμβούλιο υπ' αυτή την έννοια. Μιλήσατε για τον διορισμό του επόπτη προστασίας δεδομένων. Άκουσα όλη τη φημολογία, τη σχετική φημολογία και μπορώ να σας πω μόνο το εξής. Η διαδικασία διορισμού ε, βρίσκεται εν εξελίξη και θα πρέπει να κατανοήσετε ότι δεν μπορώ να σχολιάσω μία διαδικασία εν το γίγνεσθε. Ο επόπτης αυτή η αρχή είναι ανεξάρτητη, κάτι το οποίο κατοχυρώνεται από τις συνθήκες και γι' αυτό ακριβώς σας λέω ότι η Επιτροπή δεν επιλέγει τον επόπτη για να διασφαλιστεί αυτή η ανεξαρτησία. Άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να, δεν μπορεί να ε, έχει άποψη επί της διαδικασίας για να μην επηρεάσει την ε, όλη εξέλιξη έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης ανεξαρτησία. Εάν το ζήτημα αυτό συζητηθεί από το Διευθυντήριο, θα λάβω το λόγο και θα ταχθώ υπέρ μιας λύσης που διασφαλίζει την ανεξαρτησία και αξιοπιστία του επόπτη προστασίας προσωπικών δεδομένων. Επειδή είναι εν εξελίξη αυτή η διαδικασία, είμαι πεπισμένη ότι ο κύριος Σεφκοβιτς προωθεί το θέμα όπως πρέπει. Όπως είπε η κυρία Σαρτζεντίνη και η κυρία Σίπελ αναφέρθηκε στο εξής. Μας είπε ότι στου, σε δύσκολους καιρούς τα κράτη-μέλη δεν μας ενδιαφέρει, δεν θέλουμε να περικοπούν τα δικαιώματα, θα πρέπει να διατηρηθούν. Και ακριβώς αυτό προσπαθούμε να προβάλλουμε, ελπίζοντας ότι στα κράτη-μέλη τα σημαντικά μπορούν να προωθηθούν και τα λιγότερο σημαντικά ε, θα περικοπούν αν χρειαστεί, αν αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο. Μιλήσατε για την ελεύθερη διακίνηση και είπα και εγώ ότι αυτό είναι ένα ε, θεμελιώδες δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών και έτσι το αντιμετωπίζουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες. δείτε το ευρωβαρόμετρο. Βλέπετε τις ερωτήσεις που υποβάλλονται στον κοινό πολίτη και βλέπετε ποιες είναι και οι βασικές αξίες ε, οριζόντια που προβάλλουν οι πολίτες. Όλοι υπερασπίζονται την ελεύθερη διακίνηση Άρα πρόκειται για θεμελιώδες δικαίωμα το οποίο έτσι αντιλαμβάνονται και οι πολίτες των κρατών μελών και έχετε δίκιο. Εστιάζουμε την προσοχή μας σε ορισμένες περιφέρειες εκεί που ανακύπτουν δυσχέρειες. Γι' αυτό ζητώ από τους δημάρχους, από τις μικρότερες περιφέρειες σε αυτή τη ε, διάσκεψη, έτσι ώστε να δούμε ποιοι είναι οι κανόνες και ποιες οι δυνατότητες, καθώς και τα χρηματοδοτικά μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Διότι ακούμε πολλούς ε, μύθους και πολλές φορές είναι δύσκολο να αντιδράσουμε. Έλαβα και επιστολές από ορισμένους δημάρχους οι οποίοι καλοί την πίστη προσπαθούν να τα καταφέρουν αλλά τους κατακλείζουν τα γεγονότα γιατί δεν είναι οριζόντιο το θέμα, επικεντρώνεται σε ορισμένες περιφέρειες. Εάν το δείτε οριζόντια είναι πολύ μικρό. Δηλαδή ο αριθμός των πολιτών, των ατόμων ανακεφαλή είναι ε, πολύ μικρός, αλλά αν το δείτε σορευτικά ή τοπικά ή περιφερειακά, τότε διονγκώνεται το θέμα. Η κυρία Λάντφορντ μίλησε για το δικαίωμα της σιωπής. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα, καθώς και το τεκμήριο της αθωότητας. αποτελούν ενιαίο νομοθέτημα. Πέρα δηλαδή από τα κριτήρια του ΕΔΑΔ, δεν, δεν, υπάρχει, δεν είναι αρκετό δεν είναι αρκετή επαρκής αυτή η προστασία, διότι 11 κράτη παραβιάζουν το τεκμήριο της αθωότητας μεταξύ του, μεταξύ του 7 και του 12 στα, στην περίπτωση, σε 25 περιπτώσεις και αυτό είναι η άκρη του παγόβουνου. Γιατί ξέρετε ότι πριν φτάσει το θέμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το θέμα έχει διονγκωθεί. Και πολλές φορές Ήδη προβλέπεται η προστασία θεωρητική τουλάχιστον ως προς το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά αυτό είναι καθαρά θεωρητικό, διότι μας απασχολούν ορισμένες πτυχές του τεκμηρίου αθωότητας, αλλά δεν μπαίνουμε στην ουσία του ποινικού δικαίου σε σχέση με τις επιμέρους ευθύνες και την ε, παρουσίαση αποδεικτικών στοιχείων. Οι εμπειρογνώμονες λοιπόν έλαβαν υπόψη το common law, το βρετανικό σύστημα καθώς και το ευρωπαϊκό, το υπηρετικό σύστημα και προσπαθούν να προβάλλουν κάτι το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί. Το θέμα της Ρουμανίας, ως προς το θέμα της Ρουμανίας, και το πρόσφατο νομοθέτημα ότι δηλαδή η διαφθορά ε, δεν αποτελεί αστικό αδίκημα πλέον. Στην ε, ειδική έκθεση την οποία συντάσσουμε θα το δούμε το θέμα. τον Ιανουάριο δηλαδή θα το αντιμετωπίσουμε, αλλά βεβαίως ε, ανησυχούμε για τις ε, κακές αυτές, ε, δυσίωνες αυτές εξελίξεις στη Ρουμανία ως προς την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η κυρία Γκένς ε, ρώτησε κατά πόσο θα πρέπει να γίνει επέκταση του εντάλματος για ποινικά αδικήματα. σε σχέση με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το Κοινοβούλιο υποστήριξε την Επιτροπή επί του θέματος. Το Συμβούλιο ε, έδρασε ομόφωνα έτσι ώστε να μην δεχτεί οποιασδήποτε αλλαγές για τη διεύρυνση του πεδίου εντολής. Άρα καλύτερα να υποβάλλετε το ερώτημα στο Συμβούλιο. Ως προς το κράτος δικαίου, ξέρετε ότι αυτό αποτελεί ευθύνη του Προέδρου ε, Μπαρόζο σε συνεργασία με μένα, αλλά εκείνος αναλαμβάνει την ευθύνη και ο πρόεδρος ε, Μπαρόζο μου έλεγε ότι οι εποχές είναι κάτι το σχετικό, δηλαδή η άνοιξη έρχεται νωρίτερα σε μερικούς και αργότερα σε άλλους, ανάλογα αν βρίσκονται στο βορρά ή στο νότο. Νομίζω ότι ο κύριος Μπαρόζο λαμβάνει υπόψη την νότια προσέγγιση περί άνοιξης. Και αν τον δείτε και στους διαδρόμους πείτε του ότι θα θέλατε αυτό το κείμενο το συντομότερο δυνατόν. Νομίζω ότι είμαστε σχετικά έτοιμοι. Θα δούμε πότε θα το υποβάλει, πότε θα το υποβάλει ο πρόεδρος Μπαρόζο. Ο συνάδελφός σας Βρόνς δεν είναι παρόν, άρα δεν χρειάζεται να απαντήσω. Ως προς την κυρία Ιντβελτ, για τον οδικό χάρτη για τα δικαιώματα των ΛΟΑΔ Θα ήθελα να πω ότι εξ αρχής αυτό που κάνω εδώ και πολλά χρόνια είναι να εξασφαλίσω την συστηματική συμμόρφωση με το άρθρο, με το άρθρο 21 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και των νομοθετημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμάστε την οδηγία περί προσόντων που προβλέπει την προστασία από, σε περιπτώσεις που κανείς προβαίνει σε διώξεις, σε, σε ή μη πρόσληψη ή μη χορήγηση ε, ασύλου ε, λόγω γενετήσιου προσανατολισμού. Γι' αυτό δηλαδή οποιοδήποτε νομοθέτημά μας είναι αναλογικό και λαμβάνουμε τα μέτρα τα οποία είναι απολύτως αναγκαία. Ε, Επίσης, προωθούμε τα δικαιώματα των ΛΟΑΔ με βάση τους νόμους που βρίσκονται ήδη ισχύ ως προς την οδηγία απασχόλησης και ισότητας, όπου ε, ανοίξαμε πολλές διαδικασίες ε, για παραβίαση και έχουμε παρέμβει σε τακτά χρονικά διαστήματα με τα κράτη-μέλη όταν ε, παρακολείται το δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης. Είχαμε πολλές περιπτώσεις. και στους νέους νόμους επιτάπιος, δηλαδή ιδιοκτησιακό καθεστώς σε περίπτωση γάμου ή σε περίπτωση που συζεί ένα ζευγάρι κοινή στέγης. Όταν ε, ένα κράτος μέλος αποδέχεται ένα γάμο, ένα άλλο κράτος ε, μέλος δεν έχει το δικαίωμα να μην δεχτεί τις συνέπειες αυτής της έγγαμης σχέσης. Άρα στη συνήθιμα μας εργασία και μπορώ να αναφερθώ σε όλες τις περιπτώσεις, ε, γιατί και στη Χάγη στη διάσκεψη διαφέρθηκα σε όλες τις περιπτώσεις που έχουμε προς εξέταση, ε, συστηματικά προβάλλουμε αυτή την προσέγγιση σε όλα τα επίπεδα της ε, πολιτικής μας. Πρόσβαση στα έγγραφα. Ξέρω τις διαφορετικές ε, γνώμες μεταξύ ορισμένων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του δικού μας θεσμικού οργάνου. Δεν θα ήθελα να επέμβω αλλά θα ήθελα να πω ότι το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα λεπτό και το αφήνω στους εμπειρογνώμονες με τους οποίους ε, συνδιαλέγεστε. Η κυρία Μπάουερ μίλησε για ένα δύσκολο ζήτημα. Ακόμα και αν δεν είναι παρούσα, θα ήθελα να απαντήσω γιατί το το θέμα των παιδιών μετά από διαζύγια είναι λεπτό. Πολλές φορές οι αρμοδιότητές μας είναι περιορισμένες. Συνεργάστηκα με ορισμένους υπουργούς δικαιοσύνης σε δύσκολες διασυνοριακές περιπτώσεις στις οποίες μου επέσυραν την προσοχή και ο διάλογος στάθηκε γόνιμος αλλά σε μερικές μόνο περιπτώσεις. Το ερώτημα του κυρίου Βος, ως προς το ερώτημά του, νομίζω ότι απάντησα ήδη πριν και στο DPA και την προστασία δεδομένων. Ως προς το EPPO, επειδή ο κύριος Γιακολίνο είναι υπεύθυνο και παρόν εδώ, ε, για το θέμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας το θέμα είναι απόλυτα σαφές και ήταν σαφές για τους συντάκτες της συνθήκης. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε αν δεν υπάρχει ομοφωνία για την πρόταση. Θα πρέπει να ξέρετε ότι ορισμένα κράτη-μέλη βρίσκονται εκτός σχεδίου Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία και Ιρλανδία. Άλλα κράτη συζητούν την πρόταση. Υπάρχουν χώρες που τάχθηκαν υπέρ άλλες αναρωτιούνται τι πρέπει να κάνουν και η όλη συζήτηση θα προωθηθεί. Η ελληνική προεδρία θεωρεί μία προτεραιότητα και αυτό το ζήτημα Άρα ο Έλληνας υπουργό θα εργαστεί επί του θέματος να δούμε κατά πόσο μπορούμε να φτάσουμε σε ομοφωνία. Εάν όχι θα φτάσουμε στο επόμενο θέμα όπως προβλέπεται από το άρθρο 86 της Συνθήκης, δηλαδή ενισχυμένη συνεργασία με τουλάχιστον 9 κράτη-μέλη. Ε, είμαι πεπισμένη ότι θα έχουμε πολύ περισσότερα από 9 που θα θέλουν να προωθήσουν την ενισχυμένη συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Αντιπρόεδρε Ρέντινγκ, για την λεπτομερέστατη απάντησή σα. Η κυρία Γκόμε έχει ζητήσει το λόγο, παρακαλώ, πολύ σύντομα. Και αν θέλετε μετά μπορείτε να απαντήσετε. Κυρία Γκόμες, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, μπορείτε να μας ε, πείτε, όταν μιλάτε για την έκθεση κατά της διαφθοράς που έχει προβλήματα, μπορείτε να μας ε, πείτε τι εννοείτε, την περιμέναμε φέτος. Με συγχωρείτε, δεν είπα κάτι τέτοιο. Ε, το άκουσα όμως, λέει η κυρία Γκόμες. Η έκθεση κατά της διαφθοράς είναι αρμοδιότητα της κυρίας Μάλιμστρομ. Αυτό που με ρωτήσατε είχε να κάνει με τη Ρουμανία και την ε, νομοθεσία για την κατάργηση, διαγραφή της διαφθοράς ε, από τον κατάλογο των αστικών αδικημάτων. Αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εγώ είπα πως ναι, με ανησυχεί πολύ το ότι σε κάποια κρατημέλη η καταπολέμηση της ε, διαφθοράς δεν προχωρά όπως θα έπρεπε. Αλλά παρακαλώ δεν θέλω να πω τίποτα απολύτως για κάτι το οποίο είναι αρμοδιότητα της ε, Επιτρόπου Μάλιμστρομ. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και δεν τοποθετήθηκα γι' αυτό γιατί δεν ξέρω την άποψή της. Σας ευχαριστούμε κυρία Ρέντινγκ. Ευχαριστούμε πολύ τους συναδέλφους. Και κύριε Επίτροπε, είστε πάντα πρόσδεκτοι στην Επιτροπή μας. Τώρα, επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έδρα της ΣΕΠΟΛ. Ο Ούγκρος ε, Αρμόδιος Υπουργός βρίσκεται εδώ και νομίζω πως μπορούμε να συνεχίσουμε αμέσως. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τον Υπουργό να καθίσει και να έρθει εδώ. Παρακαλώ, όσοι θέλετε να αποχωρήσετε, αποχωρήστε και μετά ας συνεχίσουμε. Uh, Επόμενο λοιπόν σημείο στην ημερήσια διάταξη, η έδρα της ΣΕΠΟΛ της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας. Uh, as you know, does it work? As you know, is now Όπως γνωρίζετε, η ΣΕΠΟΛ αυτή τη στιγμή έχει έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όμως ανακοινώθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο ότι θα ε, κλείσει αυτός ο χώρος το 2014 και δεν επιθυμεί πλέον να έχει την έδρα της ΕΣΕΠΟΛ. Το Συμβούλιο αποφάσισε στις 8 ε, Οκτωβρίου ότι προτιμά έδρα της ΕΠΟΛ να είναι η Βουδαπέστη της Ουγγαρίας. 25 κράτη-μέλη κατέθεσαν μια νομοθετική πρόταση για αυτό. Γι' αυτό λοιπόν καλέσαμε τον κύριο Σάντορ Πίντερ, υπουργό, αρμόδιο υπουργό της Ουγγαρίας, για να μας κάνει την παρουσίαση. Ωστόσο, η αλλαγή της έδρας ε, χρειάζεται και τροποποίηση της νομοθετικής πράξης και έγκριση Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ως συνομοθέτες. Γι' αυτό λοιπόν καλέσαμε την νομική υπηρεσία για μια σύντομη παρουσίαση της νομικής γνωμοδότησης που ζήτησε η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για το θέμα αυτό και επίσης θα μας ενημερώσει η Λιθουανική Προεδρία για το τι ενέργειες κάνει το Συμβούλιο και πού βρίσκεται η κατάσταση εκεί. Και μετά τις παρουσιάσεις θα δώσω το λόγο στα μέλη, στους ευρωβουλευτές για να υποβάλουν ερωτήσεις. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πολύ που βρίσκεστε εδώ και που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Αν μου επιτρέψετε θα συνεχίσω να μιλώ στα αγγλικά ως πρόεδρος της Επιτροπής, έτσι συνηθίζεται. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να έρθω εδώ και να σας παρουσιάσω την αίτηση της Ουγγαρίας για την έδρα της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας. Θα σας κάνω λοιπόν την παρουσίασή μας και επιτρέψτε μου να κάνω μία παρουσίαση ανεξάρτητα από την επίσημη ε, παρουσίαση και την συγγραφή υποχρεώσεων. Το ως επικεφαλής της αστυνομίας 1991 ε, λάβαμε επιστολές από πολλούς συναδέλφους μου, Γάλλους, Βέλγους, Ιρλανδούς, ε, Ολλανδούς, αλλά και από την Αυστρία, την ε, Ελβετία που είναι οι γειτονικέ χώρες, μια επιστολή, επιστολές οι οποίες ε, βοήθησαν την χώρα μου να τροποποιήσει και να μεταρρυθμίσει τις αστυνομικές της δυνάμεις και το βασικότερο ζήτημα, αυτό που μας απασχόλησε, ήταν να ε, συνεχίσει να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται η προστασία των ε, διαφόρων χώρων. Και με τους συναδέλφους μου προετοιμαστήκαμε κατάλληλα και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι απαιτείται η κατάρτιση. Είπαμε δηλαδή πως ε, θα επιθυμούσαμε όλοι οι πολίτες της ε, Ένωσης να αισθάνονται ως τον ασφαλείς, ασφαλέστεροι, ώστε στην περίπτωση που θα προκύψει κάποιο πρόβλημα να γνωρίζουν ότι μπορούν να διαθέσουν τα αυτά μέτρα αστυνομικά ανά την ε, επικράτεια της Ευρώπης. Και αυτό θα πρέπει να το αισθάνονται και οι αδικοπραγούντες, οι εγκληματίες που δρούν ανά την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν θεωρήσαμε ότι η κατάθεση θα πρέπει να γίνεται με τρόπο ενιαίο, κοινό και να ακολουθούμε τις ίδιες ε, εκπαιδεύσεις ε, κατά ψυχής συνθήκες απανταχού. Δυστυχώς ε, κατά ένα διάστημα δεν μπόρεσα να επηρεάσω τη διαδικασία, αλλά τώρα που είμαι σε θέση να μπορέσω να επηρεάσω τη διαδικασία και τη λήψη αποφάσεων, αποφάσεων να, να σας κάνω λοιπόν αυτή την παρουσίαση αναφορικά με την αστυνομική εκπαίδευση και κατάρτιση. Και εμείς θέλουμε να παρέχουμε το καλύτερο, ευνοϊκότερο δυνατό κλίμα για την εκπαίδευση και την κατάσταση των νομικών. Είπαμε λοιπόν ότι αυτό που η Κομισιόν, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμούσαν ε, γιατί το 2012 τον 19 Ιουλίου εγκρίνατε, εγκρίνατε μια κοινή δήλωση με τις απαραίτητες προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρεί η έδρα των ε, ΣΕΠΟΛ. Στις 13 ε, Δεκεμβρίου οι Υπουργοί έλαβαν ε, απόφαση βάσει της οποίας ε, οι χώρες της διεύρυνσης το 2004 θα πρέπει να τύχουν ε, προτίμησης, έχουν προτεραιότητες ε, ό,τι αφορά την επιλογή αυτών των, αυτής της έδρας. Η Ουγγαρία πληρεί λοιπόν τις δηλώσεις αυτής της κοινή ανακοίνωσης Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Κομισιόν και από την προσχώρηση 2004 ξέρετε ότι καμία έδρα, καμία υπηρεσία δεν έχει ως έδρα την χώρα μου και θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε αυτά τα αντικειμενικά κριτήρια. Πρώτα απ' όλα αφορούν την εύκολη πρόσβαση, το κριτήριο 1. Το δεύτερο είναι το εξαιρετικό περιβάλλον και τα εξαιρετικά κτίρια που θα στεγάσουν αυτήν την έδρα, θέματα ε, ασυλίας ε, του προσωπικού της, ε, πολλές δυνατότητες που παρέχουμε για την εκπαίδευση των παιδιών του προσωπικού που θα στελεχώσουν την υπηρεσία και εξαιρετικές δυνατότητες σε ό,τι φορά την παροχή των υγειονομικών ε, παροχών. ε, νομίζω πως η Βουδαπέστη καλύπτει όλες αυτές τις προϋποθέσεις ε, και γι' αυτό ετούμεθα της ε, έδρας της ΣΕΠΟΛ. Επιτρέψτε μου να προσθέσω πως η ΛΕΑ δρά στην Ουγγαρία και είχαμε την δυνατότητα να συνεργαστούμε με το FBI των Ηνωμένων Πολιτειών από το 1995 όταν ξεκίνησε η συνεργασία με 28 χώρες σε επίπεδο ανώτατης δυνατή κατάρτισης για τους επικεφαλείς των αστυνομικών αρχών και για μας πρόκειται για ένα επίτευγμα για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα φιλόδοξη και υπερήφανη. Έχουμε λοιπόν αυτό το, αυτή την έδρα την Ηλέα. Βλέπουμε ότι ε, το περιοδικό Economist σε ένα δημοσίευμά του δήλωνε πως η Βουδαπέστη αποτελεί μια πόλη όπου το ε, βιωτικό επίπεδο είναι από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βρίσκεται στους 100 ε, χώρες, 100 πόλεις, συγγνώμη, βλέπετε εδώ την προσβασιμότητα Βλέπετε εδώ τους προορισμούς ε, και τις αφήξεις. Υπάρχουν περίπου 40 πτήσεις ε, ημερήσιες ε, από άλλες πρωτεύουσες. Πέντε πρωτεύουσες δεν είναι άμεσα συνδεδεμένες όπως η Λουμπλιάνα, αλλά είναι εύκολος προσβάσιμη με αυτοκινητόδρομο. Τώρα, σε ό,τι φορά την άφηξη του στο κτίριο. Είναι 22 χιλιόμετρα βρίσκεται από το αεροδρόμιο το κτίριο. Στεγάζει την έδρα και είναι εγγυημένη η πρόσβαση. Το κέντρο η έδρα λοιπόν βρίσκεται στο δυναμικό κέντρο, δυναμικό το κέντρο βρίσκεται, που συνεχώς αναπτύσσεται στο κέντρο της ε, Βουδαπέστης και να σας πω επίσης ότι εκτός από το μετρό το οποίο εξυπηρετεί το ε, Νέδρα υπάρχει και το τραμ το οποίο είναι παλιό είναι το πιο παλιό τρένο θα λέγαμε στην υπηρετική Ευρώπη από το 1916 λειτουργεί. Υπάρχουν εμπορικά κέντρα θέατρα, η όπερα βρίσκεται εγγύς του κτηρίου. Τώρα το κτίριο, το βλέπετε, είναι ένα ιστορικό κτίριο της Βουδαπέστης έχει ανακαινιστεί, έχει υπλωθεί, οι τεχνικές εγκαταστάσεις έχουν τοποθετηθεί. Υπερβαίνουμε τα κριτήρια τα οποία έχουν τεθεί για την έδρα της ΣΕΠΟΛ. 31 Αυγούστου 2014 λοιπόν θα μπορούμε να διαθέσουμε αυτό το κτίριο στην Σεπόλση του φορά τώρα τα έξοδα συντήρησης ε, του κτιρίου, ασφάλειας και όλα αυτά, το κράτος αναλαμβάνει την κάλυψη για μία δεκαετία. Δέκα χρόνια καταλαβαίνετε ότι αποτελεί με σημαντική συμβολή. Πρόκειται για 200.000 ευρώ ετησίως. Τώρα κάτι ακόμα, αν υπάρχουν δυνατότητες ε, να ασκηθεί κανείς ε, υπάρχουν ε, εγκαταστάσεις για τον ε, ελεύθερο χρόνο, να αναψυχής φυσικά, υπάρχουν ε, θέατρο, υπάρχει δυνατότητα να ακούσει κανείς μουσική, αλλά και τη δυνατότητα να ασκηθεί στο κέντρο του αθλητισμού. Μπορεί να παίξει κανείς μπάσκετ, handball, τέννις. Δυνατότητες λοιπόν ευρύτατες για επιλογή ουδήποτε θα έλεγα αθλήματος. Τώρα πέραν των, της άθλησης να αναφερθώ πως ένα ε, τμήμα του προσωπικού θα έχει διπλωματικό καθεστώς και θα παρέχουμε τις ε, απαραίτητες ασυλίες κλπ. Τώρα, μια βασική ερώτηση, τι θα γίνει με τις οικογένειες των ε, υπαλλήλων. Υπάρχουν πολλά σχολιά, ιδιωτικά, δημόσια. Βλέπετε λοιπόν εδώ τις αριστερά τη στήλη διάφορες ηλικίες, και τις ε, γλώσσες ε, αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ισπανικά από την ηλικία των τριών ετών ε, γίνεται δασκαλία σε αυτές τις τέσσερις γλώσσες για έναν αρκετά σημαντικό αριθμό μαθητών και μετά μπορεί να στοιχήσουν τις σπουδές στα γαλλικά, γερμανικά, αγγλικά Τώρα, σε ό,τι φορά την υγειονομική περίθαλψη, έχετε σε μερικά χιλιόμετρα ε, νοσοκομείο το οποίο μπορεί να σας ε, παράσχει τις ε, απαραίτητες θεραπείες Επίσης υπάρχει δυνατότητα να εργαστούν ε, τα παιδιά, οι σύζυγοι σε κοντινή απόσταση και είναι πολύ εύκολη πρόσβαση. Τώρα, με λίγα λόγια να πω ότι ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις προσδοκίες του Συμβουλίου των Υπουργών, στις προσδοκίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και στις προσδοκίες της ε, Κομισιόν. Δεν υπάρχει κάποια υπηρεσία της Ένωσης που να έχει την έδρα της στην Ουγγαρία και να σας πω ότι ο Σπουλυπουργών ομοφόνος ε, εκφράστηκε υπέρ της υποψηφιότητάς μας. Και τώρα να σας δείξω πώς έχουμε τροποποιήσει, πώς μετατρέψαμε μάλλον αυτό το κτίριο σε λίγο χρονικό διάστημα για να παρέχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις ε, ως έδρα της ΕΠΟΛ. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι πρόθυμος να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Akkor eh, köszönöm eh, Λοιπόν, για μια ακόμα φορά σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Υπουργό για την παρέμβασή του και θα πρέπει να δώσουμε ευκαιρία στα μέλη να θέσουν ερωτήσεις επειδή χρειάζεται να αποχωρήσει στις 5 θα ανοίξω τώρα τη ε, δυνατότητα στις έρωτα αποκρίσεις έχω στον κατάλογο μου τον κύριο Γκόνς Mrs. Bauer, Mr. Tavares? Okay. Then uh, uh Ευχαριστώ. Να συγχαρώ τον Υπουργό για την παρουσίασή του και την πρότασή του. Είναι εξαιρετική παρουσιάζονται όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που η Βουδαπέστη προσφέρει για μία από τις ε, υπηρεσίες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, ρωτώ το θέμα της πολιτικής στήριξης πίσω από την πρότασή σας. Ακούσαμε διάφορα αντιευρωπαϊκά ευρωπαϊκές δηλώσεις ε, ο οποίος δηλώνει ο Πρωθυπουργός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εχθρός της Ουγγαρίας. Και τώρα βλέπω ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να προσελκύσετε αυτήν την έδρα. Ελπίζω να το πετύχετε, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω αυτού του είδους την αντίφαση. Δεν ξέρω πώς μπορείτε να συμβιβάσετε και να συνδυάσετε αυτές τις δύο θέσεις. Να αναφέρω επίσης πως μπορεί να ακούσατε κάποιες από τις ανησυχίες που εκφράστηκαν εδώ στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και που αφορούσαν τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου Αναφέρθηκε επίσης ότι θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον είναι η βέλτιστη των αποφάσεων αυτή να δημιουργηθεί στην ε, Βουδαπέστη η έδρα της ΣΕΠΟΛ. Ελπίζω λοιπόν με την νέα κυβέρνηση τα πράγματα να πάνε καλύτερα και ότι η απόφαση αυτή να μην είναι βράχη πρόθεσμη αλλά μακρόπνοη η νομική υπηρεσία uh, uh, η νομική υπηρεσία θα μιλήσει αργότερα είναι χωριστό θέμα αλλά θα ήθελα να αναφέρω ότι με απασχολεί η όλη διαδικασία πως λήφθη η απόφαση στο Συμβούλιο δεν είναι πλάκι ούτε το Κοινοβούλιο ούτε η Κομισιόν αλλά αυτό είναι διαφορετικό θέμα το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε αργότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα την... Ε, μάλλον θα ήθελα να λάβω το λόγο αφού ακούσω την θέση της νομικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου. Θα πω προς τον στον κύριο Υπουργό, τον ευχαριστώ για την παρουσίαση και για την ενημέρωση, αλλά εγώ έχω ισχυρέ επιφυλάξει σχετικά με την διαδικασία που ακολουθήθηκε. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ακούσω πρώτα την νομική υπηρεσία και καλώ ήρθατε κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για την παρουσίασή σας. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστερημένη αφεξή μου, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να κάνω πολλά πράγματα, μια ψηφοφορία για παράδειγμα, σε μια άλλη επιτροπή. Μια ερώτηση επί της διαδικασίας. Ε, πώς βλέπετε εσείς τη διαδικασία, διότι αν κατάλαβα καλά, είναι μια πρόταση αυτή που ήρθατε και μας παρουσιάσατε. Δεν έχει ληφθεί η οριστική απόφαση. Γι' αυτό λοιπόν σας ερωτώ σε ποιο στάδιο της απόφασης βρισκόμαστε, σε ποιο στάδιο της διαδικασίας. διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μπάουερ, ο κύριος Ταβάρες. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αναφερθώ και εγώ στην διαδικασία που θα ληφθεί έτσι ώστε να αποφασιστεί ποια θα είναι η έδρα της ΕΣΕΠΟΛ. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω πρώτα να ακούσουμε την άποψη της νομικής υπηρεσίας και έπειτα να σχολιάσουμε. Γι' αυτό λοιπόν προσωπικά θα περιμένω μέχρι να ακούσω την νομική υπηρεσία. Όμως μπορώ να σας πω ότι σήμερα μιλώ και ως σκιώδης εισηγητής για το φάκελο της Ευρωπόλ και ως εισηγητής για την έκθεση, το ψήφισμα πλέον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του κράτους δικαίου και την προστασία των πολιτών στην Ουγγαρία. Να σας πω ότι είναι δύσκολη η θέση μου. Θα ακούσουμε και την άποψη της νομικής υπηρεσίας σε λίγο, όμως το γεγονός είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα τις ε, αποφάσεις του για το φάκελο της Ευρωπόλη. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συγχωνευτεί Ευρωπόλη και ΣΕΠΟΛ ε, είναι κάτι που με βρίσκει αντίθετο, με έβρισκε ανέκαθεν αντίθετο και εμένα και την ομάδα μου. Και κάτι τέτοιο θα είχε και επιπτώσεις. Όμως να πω πως ε, καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ για την μεταφορά της έδρας της πόλης στη Βουδαπέστη. Είναι πολύ όμορφη πόλη η Βουδαπέστη. Όμως τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ως έργο να, τη διασφάλιση της καλής συνεργασίας. Και τώρα έχει ήδη αρχίσει μια νομοθετική διαδικασία. Το Συμβούλιο ήταν ε, στο ίδιο μήκο κύματο με το Κοινοβούλιο, όμως πρέπει να ακολουθήσουμε κάποιους ε, κανόνες, νομικούς κανόνες και πρέπει λοιπόν να περιμένουμε πρώτα να ολοκληρωθεί η νομική διαδικασία πρωτού περάσουμε σε κάποια άλλη. Εσείς ε, δεν πιστεύετε ότι μπορεί να διακυβευτεί το αποτέλεσμα της απόφασης δεδομένου ότι η απόφαση που ελήφθη στο Συμβούλιο δεν ήταν νομικά επαρκής. Εσείς δεν θεωρείτε πως παρεκκλίνεται από την νομική διάσταση της πρότασης αυτής. Έπειτα, δεν συμφωνείτε ότι και το Κοινοβούλιο πρέπει να συναποφασίσει για το θέμα αυτό, για την έδρα της ΣΕΠΟΛ. Τώρα, δεν θα αναφερθώ σε όλες τις λεπτομέρειες της έκθεσης σχετικά με το καρτός και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ουγγαρία, όμως ένα σημείο έχει τραβήξει την προσοχή μας. Όταν μιλάμε για αστυνομική συνεργασία, και την έδρα λοιπόν της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας που θα πάει στη Βουδαπέστη. Μιλάμε για μια έκθεση που δεν ε, είναι δική μας αλλά των Ηνωμένων Εθνών. Η κυρία Ναβή Πιλάη, αρμόδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχει αποφανθεί ότι ότι η καταπάτηση των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων από την αστυνομία στην Ουγγαρία είναι έντονη και θα ήθελα λοιπόν να ακούσω την άποψή σας όσον αφορά τις ε, ενέργειες της αστυνομίας και όσο και εσείς πείτε μου θεωρείτε ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση σε σχέση με την έκθεση αυτή των Ηνωμένων Αθηνών. Και εάν έχει βελτιωθεί η κατάσταση, Πώ σκοπεύετε να προχωρήσετε και αν δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση, τι σκοπεύετε να κάνετε για να γίνει αυτό. Διότι η έδρα της ΕΠΟΛ στην Βουδαπέστη είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θα μπορούσατε να το χρησιμοποιήσετε ως αφορμή για να βελτιωθεί η κατάσταση με την αστυνομία και τις επιθέσεις της αστυνομίας στις μειονότητες. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ταβάρες. Όπως ε, ακούσατε, μετά την απάντηση του Υπουργού θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τη νομική υπηρεσία. Ναι, η δική μου παρέμβαση, λέει ο κύριος Ταβάρες, είχε ακριβώς να κάνει με, το, με αυτά που θα ακούσουμε από την νομική υπηρεσία, διότι δεν μπορούμε να ακούσουμε την απάντηση του Υπουργού πριν, ε, αν δεν έχουμε πρώτερα ενημερωθεί από τη νομική υπηρεσία. Ας δώσουμε πρώτα το λόγο στον Υπουργό να απαντήσει στις ε, ερωτήσεις. Προτείνω μετά θα ακούσουμε την νομική υπηρεσία και έτσι καλλιώς δεν μας λείπουν οι ερωτήσεις. Ο συνάδελφος Δίας Δεμέρα είπε πριν ότι θα ρωτήσει απευθεία την ε, νομική υπηρεσία και όπως σας είπα μετά θα λάβει το λόγο και εκπρόσωπος της Λιθουανικής Προεδρίας. και θα τοποθετηθεί σε ζητήματα Προεδρίας και Συμβουλίου. Γι' αυτό λοιπόν ας αφήσουμε πρώτα τον Υπουργό να απαντήσει, αν συμφωνείτε και μετά όλα τα υπόλοιπα. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Άκουσα τις ερωτήσεις σας με προσοχή και να σας πω ότι χαίρομαι. Χαίρομαι γιατί καμία από τις ερωτήσεις δεν είχε εκφράσει αμφιβολίες για το αν είναι κατάλληλη η πόλη Βουδαπέστη για την έδρα της ΕΠΟΛ. Κανείς δεν είχε την άποψη ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την μετεγκατάσταση της ΕΠΟΛ στην Ουγγαρία. Υπάρχει λοιπόν η συμφωνία, ομοφωνία, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις από την Βουδαπέστη για τη μεταφορά της έδρας της Επολεκή. Τώρα όμως θα αρχίσω απαντώντας την κυρία Γκέντς. Με ρωτήσατε εάν υπάρχει πολιτική στήριξη στον Υπουργό Εσωτερικών. Μπορώ να σας πω πως ναι. Εγώ προσωπικά απολαμβάνω την πολιτική στήριξη όλων των βουλευτών και των εξοκοινευουλευτικών κομμάτων όσον αφορά την ε, ΣΕΠΟΛ. Όλοι οι πολίτες της Ευρώπης επιθυμούν να απολαμβάνουν την καλύτερη δυνατή αστυνομική προστασία. Έχουμε λοιπόν τους ίδιους στόχους, θέλουμε να αισθανόμαστε ασφάλεια στην Ευρώπη, σε όλα τα κράτη-μέλη και αυτό θα συμβεί μόνο εάν η αστυνομία σε όλα τα κράτη-μέλη έχει την ίδια κατάρτιση. Αυτό είναι κάτι στο οποίο συμφωνούν ομόφωνα όλοι, ανεξάρτητα από πολιτική τοποθέτηση. Γι' αυτό λοιπόν μπορώ να σας πω ότι έχω 100% ε, τη στήριξη του Κοινοβουλίου. Και η παρουσίαση αυτή σας έδειξε ότι υπάρχει ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί πάρα πολύ καλά και κανείς δεν αμφισβήτησε την ε, ορθή λειτουργία της αστυνομίας στην Ουγγαρία. Και να σας παραπέμψω και σε μια δημοσκόπηση που έγινε πριν από λίγες μέρες, σύμφωνα με την οποία όταν ερωτήθηκαν οι Ούγγροι πολίτες για το για το ποιος τομέας ε, απολαμβάνει την ε, μέγιστη εμπιστοσύνη τους, απάντησαν σε πρώτη θέση η Ακαδημία Επιστημών και σε δεύτερη θέση την Ουγγρική Αστυνομία. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι το έργο μας είναι πολύ καλό και γι' αυτό έχουμε λάβει και την υποστήριξη των περισσότερων κρατών μελών. Να προσθέσω επίσης ότι το Υπουργείο Εσωτερικών της Ουγγαρίας έχει επεκτείνει τις αρμοδιότητες του, έχει αλλάξει ο ποινικό κώδικας μέσα σε ένα χρόνο, έχουν εισαχθεί νέα δικονομικά δικαιώματα και αυτά είναι εναρμονισμένα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και πραγματικά η Ουγγρική δικαιοσύνη έχει πολύ υψηλό επίπεδο κατάρτισης και λειτουργίας. Είναι μία αλυσίδα η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και στο τέλος αυτής ή στην αρχή αυτής είναι και η κατάρτιση των αστυνομικών. Τώρα, υπάρχουν κάποιες αρχές για τις οποίες έχουν συμφωνήσει όλοι στο Συμβούλιο. για την ΣΕΠΟΛ. Να σας πω ότι η υποψηφιότητά μας έχει προχωρήσει αρκετά. Έχει οριστεί η Βουδαπέστη ως επίσημη υποψήφια πόλη και δεν έχει αποφασίσει το Συμβούλιο κάτι από μόνο του. Το Συμβούλιο αυτό που αποφάσισε είναι ότι η Ουγγαρία είναι μια χώρα την οποία μπορεί να υποστηρίξει απόλυτα για να φιλοξενήσει την έδρα της ΕΠΟΛ και τώρα χρειαζόμαστε την στήριξη και την σύμφωνη γνώμη και την δική σας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα κύριε Τάβαρες. μας ε, ρωτήσατε αν συναποφασίζει και το Κοινοβούλιο. Φυσικά, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου δεν ισχύει καμία απόφαση του Συμβουλίου. Δεν γνωρίζω αν έχει ήδη αποφανθεί το Κοινοβούλιο, αν έχει ήδη αποφασίσει γι' αυτόν υπάρχει κάποια γνωμοδότηση κατά τη διάρκεια των ε, προετοιμασιών μου μου είπαν ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα οριστικά το Κοινοβούλιο και εδώ ότι δεν θέλει να βιαστεί στη λήψη απόφασης και πώς θα περιμένει να πληροφορηθεί την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρώτα. Τώρα, από πολιτική σκοπιά, δεν τίθεται θέμα εάν είναι όλα εντάξει. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες τις οποίες θα επεξεργαστούμε, αλλά να πω κάτι για την έκθεση των Ηνωμένων Εθνών και για τις επιθέσεις της αστυνομίας ε, κατά των μειονοτήτων. Να σας πω ότι στην Ουγγαρία έχουμε δυσκολίες, έχουμε προβλήματα με τους Ρωμά, με την μειονότητα των Ρωμά. Το 2010 και το 2011, όταν ανέλαβα την ε, θέση αυτή στο Υπουργείο Εσωτερικών, είχαμε σοβαρά προβλήματα και ενδεχομένως τα προβλήματα που προέκυψαν με τους Ρωμά η αστυνομία να μην αντέδρασε έτσι όπως θα έπρεπε. Το θέμα όμως αυτό το αντιμετωπίσαμε με κατάρτιση. Είχαμε κατάρτιση, είχαμε καλέσει συναδέλφους ε, για να υποβάλουν προτάσεις κατάρτισης και είχαμε λοιπόν ένα σχέδιο που προτάθηκε από συναδέλφους Σουηδούς και Δανούς για την κατάρτιση των αστυνομικών δυνάμεων αλλά και για κατάρτιση της ε, τοπικής αυτοδιοίκησης και όλων των ε, αρμόδιων φορέων. Και χάρη σε αυτά τα μέτρα κατάρτισης δεν έχουμε πλέον τέτοια προβλήματα και τέτοιες επιθέσεις στις μειονότητες. Επίσης να σας πω ότι η Ουγγαρία έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Οι μειονότητες εκεί έχουν το δικαίωμα να ε, συστήνουν τα δικά τους ε, συμβούλια, γνωμοδοτικά συμβούλια, τις ε, δικές του είναι κάπως αυτόνομες. και σε περίπτωση προβλημάτων απευθυνόμαστε στους εκπροσώπους των μειονοτήτων αυτών για την επίλυση των προβλημάτων. Και πρέπει να πω ότι τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί ιδιαίτερη πρόοδος στον τομέα αυτό της συνεργασίας. Νομίζω πως απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις σας, μόνο κάτι επί της διαδικασίας. Να σας πω ότι 25 κράτη-μέλη στηρίζουν αυτή την πρόταση που υπέβαλε το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε λοιπόν 25 κράτη-μέλη που στηρίζουν την υποψηφιότητά μας. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, τότε θα ήθελα να απευθυνθώ στην νομική υπηρεσία για να μας παρουσιάσει την γνωμοδότησή της που ζήτησε η Επιτροπή μας για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον Υπουργό για την παρουσίασή του, για την παρουσίαση της ε, Ουγγρικής υποψηφιότητας για την έδρα της ΕΠΟΛ. Γνωρίζω πως πρέπει να φύγετε στις 5. Γι' αυτό λοιπόν σας επιτρέπουμε να φύγετε. Μόλις με ενημέρωσε η γραμματεία ότι πρέπει έτσι καλλιώς να φύγετε. Παρακαλώ λοιπόν, νομική υπηρεσία, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Thank you, Chair. <clears throat> In November we... Το Νοέμβριο λάβαμε ένα αίτημα από εσά για να γνωμοδοτήσουμε νομικά σχετικά με τη νομική βάση και την διαδικασία λήψη αποφάσεων που χρειάζεται για την αλλαγή της έδρα τη Ευρωπαϊκή Αστυνομικής Ακαδημίας. Υπήρξαν πολλές ερωτήσεις και θα προσπαθήσω λοιπόν σύντομα να σας παρουσιάσω τις απαντήσεις και τα κύρια συμπεράσματά μας. Η πρώτη ερώτηση είχε να κάνει με το εάν από την ε, στιγμή της θέσης ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας και έπειτα η συνήθις νομοθετική διαδικασία είναι η κατάλληλη διαδικασία για την ε, ανάμειξη του Κοινοβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση της απόφασης πόλη. Το συμπέρασμά μας είναι ότι από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας, η σωστή νομική βάση για την τροποποίηση της απόφασης σχετικά με τη ΣΕΠΟΛ είναι το άρθρο 87 παράγραφος 2b λατινικό της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι μια διάταξη η οποία αντικατέστησε το άρθρο 30 της πρώην συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ήταν τότε η νομική βάση για την απόφαση της ΕΠΟΛ. Το άρθρο 87 παράγραφος 2b δίνει τη δυνατότητα χρήσης της συνήθως νομοθετικής διαδικασίας. Η δεύτερη ερώτηση ήταν, αποτελούνταν μάλλον από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος έχει ως εξής, εάν η διαδικασία λήψης αποφάσεων πρέπει πλέον να είναι διαφορετική, δεδομένου ότι η τροποποίηση για την απόφαση της ΕΠΟΛΑ αφορά την έδρα της. Η απάντηση είναι όχι. Ο μόνος τρόπος για να τροποποιηθεί το άρθρο 4 της απόφασης ΣΕΠΟΛ είναι μέσω της συνήθως νομοθετικής διαδικασίας. Δεύτερο σκέλος της ερώτησης είναι εάν το άρθρο 341 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μπορεί να εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το άρθρο 341 αφορά τον ορισμό της έδρας των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Η ΣΕΠΟΛ δεν είναι ένα θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως αποτέλεσμα το άρθρο 341 δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωση αυτή. Η ΣΕΠΟΛ είναι ένα σώμα, απλά ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τρίτη ερώτηση αφορούσε την, ε, το νομικό καθεστώς της κοινή ευρωπαϊκής προσέγγισης για τις ε, αποκεντρωμένες υπηρεσίες και οργανισμούς και αν αυτό έχει νομικές επιπτώσεις στη διαδικασία τροποποίησης της απόφασης ΕΠΟΛ. Η παράγραφος 5 της Κοινής Εδήλωσης Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Κομισιών για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες καταδεικνύει ξεκάθαρα ότι και η κοινή δήλωση και η κοινή προσέγγιση έχουν νομικά μη δεσμευτικό χαρακτήρα και είναι με επιφύλαξη οι κατάλληλε διαδικασίε στην ε, νομοθετική διαδικασία. Επομένω, το έγγραφο αυτό δεν έχει νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα και δεν ε, επιβάλλει νομική υποχρέωση στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα στην ε, νομοθεσία. Τα θεσμικά όργανα έχουν δεσμευτεί να λάβουν υπόψη την κοινή προσέγγιση στα πλαίσια των μελλοντικών τους αποφάσεων σχετικά με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η κοινή προσέγγιση έχει οποιασδήποτε νομικά δεσμευτικές επιπτώσεις στην νομοθεσία και την νομοθετική διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την τροποποίηση του άρθρου 4 της απόφασης ΣΕΠΟΛ. Τέταρτη ερώτηση. Το βάρος και οι συνέπειες της πολιτικής απόφασης μιας προσωρινής μεταγκατάστασης της έδρας της ΕΠΟΛ που ελήφθη κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 8 η Οκτωβρίου 2013. Λοιπόν, μια αλλαγή τη έδρας τη ΕΠΟΛ θα απαιτεί είτε τροποποίηση της απόφασης ΕΠΟΛ, είτε μια νέα νομοθετική πράξη που θα ανακαλεί την απόφαση ΕΠΟΛ. Και οι δύο επιλογές απαιτούν τη χρήση διατάξεων τη συνθήκη που ισχύει αυτή τη στιγμή. Στην περίπτωση της ΕΠΟΛ μιλάμε για τα άρθρα 87 παραγραφο 2 2b, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις για τη χρήση της συνήθης νομοθετικής διαδικασίας και θεωρεί το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συνομοθέτες. Η πολιτική απόφαση που ελήφθη κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων δεν μπορεί να οδηγήσει σε παρέκκληση από την ε, διαδικασία λήψης αποφάσεων όπως προβλέπεται από τις συνθήκες, ούτε να έχει δεσμευτική ισχύ για το Κοινοβούλιο. Και η προσωρινή φύση μιας νομοθετικής ε, πράξης δεν έχει επιπτώσει στη διαδικασία έγκρισης ή τροποποίησης της πράξης, κάτι το οποίο ε, αναφέρεται και στις συνθήκες. Ε, συμπερασματικά, η μετακίνηση της έδρας της ΕΠΟΛ στη Βουδαπέστη, ακόμα και, ως, ε, και με προσωρινό χαρακτήρα, είναι νομικά μόνο μια πολιτική συμφωνία. Και η πολιτική αυτή συμφωνία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τα θεσμικά όργανα. Δεν μπορεί όμως να ανακαλέσει τα προνόμια και τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου στη συνήθινη νομοθετική διαδικασία. Η πέμπτη ερώτηση τώρα αφορούσε τη σχέση ανάμεσα στην πρόταση για κανονισμό της Ευρωπόλ και την ε, πιθανή νομοθετική πρωτοβουλία κάτω από το άρθρο 76 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αλλαγή της έδρας της ΕΠΟΛ. Το άρθρο 76 αναφέρει ότι η συνεργασία σε δικαστικά και ποινικά ζητήματα και αστυνομική συνεργασία μπορεί να βασιστεί είτε σε πρόταση της Κομισιόν είτε σε πρωτοβουλία ε, από το 1 τέταρτο τουλάχιστον των κρατών μελών. Και στην συγκεκριμένη περίπτωση η πρωτοβουλία των κρατών μελών κατά από το άρθρο 76 είχε τη μορφή πρότασης τροποποίησης της απόφασης ΣΕΠΟΛ. Ως ότου ανακληθεί η απόφαση της Επόλ παραμένει Μία νομοθετική πράξη σε ισχύ. Είναι λοιπόν δυνατόν να τροποποιηθεί αυτή, ακόμα και αν υπάρχει πρόταση που συζητιέται και γίνονται διαπραγματεύσεις οι οποίες ενδεχομένως οδηγήσουν σε ανάκληση της απόφασης σε πόλ, όπως η πρόταση για τον κανονισμό Ευρωπόλ. Τώρα, για το αν το, τα προνόμια του Κοινοβουλίου υπονομεύονται στην περίπτωση πρωτοβουλίας, ε, σύμφωνα με το άρθρο 76, σε περίπτωση τέτοιας λοιπόν πρωτοβουλίας ε, με την ε, μορφή πρότασης τροποποίησης του, της απόφασης ΕΠΟΛ, η απάντηση έχει ω εξή. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα πρέπει να είναι η συνήθι νομοθετική διαδικασία. Εάν η αρχική πρόταση είναι μια πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή μια πρωτοβουλία κρατών μελών, δεν έχει καμία απολύτως ε, συνέπεια στην ε, εφαρμοστέα νομοθετική διαδικασία, η οποία καμια απολυτω συνεπεια στην εφαρμοστεα νομοθετικη ίδια και στι δύο περιπτώσει. Επομένω. Στην περίπτωση πρωτοβουλίας υπό το άρθρο 76 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα προνόμια του Κοινοβουλίου δεν θα υπονομευθούν. Μία τέτοια πρωτοβουλία θα απαιτεί τη χρήση της συνήθι νομοθετικής διαδικασίας για την έγκριση της νομικής πράξης, το οποίο σημαίνει ότι θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία όπως εκείνη που θα ακολουθηθεί για την έγκριση του κανονισμού Ευρωπόλ. Αυτά ήταν ε, εν συντομία τα συμπεράσματα της ανομικής μας εγγνωμοδότησης και αν έχετε ερωτήσεις με χαρά να τις απαντήσω. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και συνάδελφοι. Uh, συνάδελφοι, θέλουμε να ακούσουμε αμέσως τη Λιθουανική Προεδρία θέλετε να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας τώρα άμεσα και μετά να ακούσετε τη Λιθουανική Προεδρία. Πρώτα την ακούμε λοιπόν και μετά υποβάλλουμε τις ερωτήσεις. Θα ήθελα να λάβει το λόγο η Προεδρία. Okay. Uh, good uh. Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, αγαπητά μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και προσκεκλημένοι. Χαίρομαι ιδιαίτερα που με αυτή την ευκαιρία μπορώ να ε, υπογραμμίσω τη θέση της Προεδρίας όταν αναλάβαμε αυτό το επιπλέον εγχείρημα, το οποίο δεν ήταν αρχικά προγραμματισμένο για την Προεδρία μας. Όμως αναγκαστήκαμε να βρούμε μία κατεπίγουσα λύση. Σας ευχαριστώ πολύ για την εκτενή σας επεξήγηση, την επεξήγηση της νομικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου που αντικατοπτρίζει τη θέση μας όταν αναλάβαμε αυτό το εγχείρημα. Όλοι γνωρίζουμε ότι η επίλυση του ζητήματος αυτού έπρεπε να προωθηθεί εξαιτίας της μονομερούς απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου να μην ε, δεχτεί να φιλοξενήσει στο Μπραμσχιλ την ε, ΣΕΠΟΛ και τον Ιούνιο το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων από κοινού με τη ΛΥΜΠΕ ασχολήθηκε με το θέμα και θεώρησε ότι το σχέδιο κανονισμού της Europol όπου άρχισε, με το οποίο άρχισε η συγχώνευση ε, τη ΣΥΠΟΛ με το Europol δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή. Υπό τις συνθήκες αυτές και αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι λίγη η τρέχουσα πολιτική θητεία και επίκυνται εκλογές, είμαστε αναγκασμένοι να εξεύρουμε σύντομα μία απλή λύση. Τον Οκτώβριο, όπως αναφέρθηκε πολλές φορές, το Συμβούλιο έλαβε ομόφωνα την απόφαση όταν απομακρυνθεί από το Μπράμσχιλ η Σίπολ να φιλοξενηθεί στη Βουδαπέστη. 25 κράτη-μέλη το δέχτηκαν αυτό. Υπέβαλαν λοιπόν μία πρόταση νομοθετικού περιεχομένου τροποποιώντας το άρθρο 4 της απόφασης για την ΣΥΠΟΛ όπου αναφερόταν ότι η έδρα της ΣΥΠΟΛ βρίσκεται στο Μπράμσχιλ. Το κείμενο αυτό προωθήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και στα Εθνικά Κοινοβούλια και αυτό έγινε στις 4 Δεκεμβρίου. Ο προτινόμενο, προτινόμενος κανονισμός θα πρέπει να εγκριθεί με συναπόφαση μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, όπως πολύ σωστά τόνισε η νομική υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα νέα κτίρια στη Βουδαπέστη θα είναι διαθέσιμα την επόμενη χρονιά στις 31 Αυγούστου και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ε, έχει παρατείνει το ομίσθωμα μέχρι το Σεπτέμβριο, θα πρέπει να εγκριθεί ο κανονισμός πριν από τις ευρωεκλογές, δηλαδή μέχρι του χρόνου τον Απρίλιο. Έτσι ώστε να γίνει η κίνηση αυτή το καλοκαίρι. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά ελπίζω οι συνομοθέτες, καθώς και εμείς στο Συμβούλιο, θεωρούμε αυτό ε, ως ένα σύνηθες εγχείρημα. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να επέλθει συμφωνία, γιατί είναι προς κοινό συμφέρον μας η ΣΥΠΟΛ να, να συνεχίσει τις εργασίες της χωρίς διακοπή και να μην υπάρχει ανασφάλεια για το προσωπικό. Ο διευθυντής της ΣΥΠΟΛ μπορεί να το ε, τονίσει αυτό να το υπογραμμίσει. Ο εισηγητής έχει ήδη διοριστεί. Από πλευρά Συμβουλίου τα κράτη-μέλη κλήθηκαν να υποβάλουν γραπτά σχόλια ως προς το κείμενο τώρα το οποίο θα συζητηθεί στις 10 Ιανουαρίου, ε, μετά δηλαδή τις χριστουγεννιάτικες διακοπές, το κείμενο αυτό θα προωθηθεί όπως είπα και πιστεύω ότι και η επερχόμενη ελληνική προεδρία θα προωθήσει το όλο θέμα μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαστε διατεθειμένοι να προωθήσουμε περαιτέρω διαπραγματεύσεις με βάση την νομική διαδικασία που προευλήθη από την ε, νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν έχετε ερωτήσεις, ευχαριστώ να απαντήσω. Θα ήθελα τώρα η Επιτροπή ενδεχομένως να παρέμβει. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω την ουσία της, του αιτήματο της Ουγγαρίας που παρουσίασε ο Υπουργός διεξοδικά. Θα ήθελα να σταθώ στην όλη διαδικασία γύρω από τις πρωτοβουλίες των κρατών μελών που ανέφεραν και οι προλαλήσαντες. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής βρίσκονται στη διαδικασία προετοιμασίας της επίσημης γνωμοδότησης της Επιτροπής ως προς αυτή την πρωτοβουλία των κρατών μελών. Μπορώ να πω τα εξής ε, με βάση αυτή την εκκρεμότητα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το σχέδιο κανονισμού που τροποποιεί την απόφαση ΣΥΠΟΛ του Συμβουλίου δεν αναφέρεται στην προσωρινή νέα έδρα του οργανισμού, όπως τόνισε και ο κύριος Ταβάρες θα θυμόσαστε ότι έχουμε επιτάπητος μία πρόταση για κανονισμό λειτουργίας της Europol που οι συνομοθέτες τώρα εξετάζουν. Όπως ανέφερε η Επιτροπή στη συνάντηση της Επιτροπής της 17 Οκτωβρίου, η πρότασή μας για τον κανονισμό της Europol υποβλήθηκε για να ασχοληθούμε διεξοδικά με την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας αστυνομικών αρχών και κατάρτισης. Ο στόχος ήταν διτός να υπάρχουν λειτουργικές συνέργειες από τη μία πλευρά, αλλά και εξοικονομήσεις από την άλλη. Και αυτό συμφαντίζοντας με τον ε, συνολικό στόχο της μεταρρύθμισης και τη σύσταση περί αποκεντρωμένων οργανισμών που ενέκριναν οι τρεις, ε, τα τρία ε, θεσμικά όργανα. Γι' αυτό θεωρούμε ότι το θέμα της έδρας της ΣΥΠΟΛ δεν θα πρέπει να ειδωθεί μεμονωμένα. Αντίθετα, θα πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη τη βάση του κανονισμού της Europol. Συνεπώς, η πρωτοβουλία των κρατών μελών για την έδρα της ΣΥΠΟΛ θα αποτιμηθεί από την Επιτροπή υπό το φως των δύο στόχων που προανέφερα. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, δύο συνάδελφοι θέλουν να παρεύουν. Δία ε, Δεμέρα, τα Βάρσα και η κυρία Αγγέντς. Ο κύριος Δία Δεμέρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στις 8 του μήνα ε, έκανα ορισμένα σχόλια τα οποία επιβεβαιώνονται όλες οι ανησυχίες και οι αμφιβολίες ε, τονίζονται και επιβεβαιώνονται σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την τεχνική εργασία της νομικής υπηρεσίας, να συγχαρώ την νομική υπηρεσία ε, η οποία με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Εμείς δεν θέλουμε να μπούμε στα χωράφια του Συμβουλίου. Δεν θα θέλαμε όμως το Συμβούλιο να κάνει το αντίστροφο. Τώρα θα ήθελα να ε, με διέπει ένα επικοδομητικό πνεύμα μέσα στα πλαίσια της ε, διαθεσμικής συνένεσης για να επιλύσουμε αυτό το θέμα. Όπως ε, είχα ήδη πει, η διαδικασία αυτή θα πρέπει να διέπεται από το άρθρο 87 ε, ε, καλωσορίσατε στο κλαμπ ε, της συναπόφασης, θέλω να πω, στο Συμβούλιο. Η ΣΕΠΟΛ δεν είναι ε, ένας οργανισμός ε, αυτού του τύπου. Μας διέπει το άρθρο 13 της συνθήκης και δεν διέπεται, δεν διέπονται οι οργανισμοί από κανένα άλλο άρθρο. Όπως είπε ε, και η νομική υπηρεσία δεν είναι δεσμευτικό το κείμενο. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην ίδια χώρα βρίσκεται και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός καινοτομία και Τεχνολογίας. Στο πέμπτο κεφάλαιο της, ε, της Συνθήκης Περιλειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Η πολιτική συμφωνία του Συμβουλίου, και αυτό το έχουμε γραπτός και το λένε και οι νομικές υπηρεσίες, η συμφωνία αυτή του Συμβουλίου δεν έχει νομικές επιπτώσεις. Η νομοθετική διαδικασία θα πρέπει να ε, βασιστεί στα προνόμια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ίδιο αφορά και το άρθρο 76. Δηλαδή μιλάμε για την τακτική νομοθετική διαδικασία. Σημερίζομαι και σημερίστηκα εξ αρχής αυτή την αρχή. Θα πρέπει να είμαστε συνεπείς. Εγώ συμφωνώ με την Επιτροπή που προώθησε μία πρόταση νομοθετικού περιεχομένου. Μέσα στα πλαίσια της σωστής λοιπόν δικαιοδοσίας θα πρέπει να προβάλλει μία νέα με βάση τις αρμοδιότητές της. Διότι και η ίδια η έκθεση, η νομική έκθεση μιλά για το εξής. Είναι δυνατόν να αλλάξει η λειτουργία της ΣΕΠΟΛ και η έδρα της με βάση μια διαδικασία εξαίρεσης. Αν και η Επιτροπή υπέβαλε μια πρόταση η οποία εάν εγκριθεί θα μπορούσε να οδηγήσει στο να γίνει παρέκκληση από την αρχική απόφαση για την ΣΕΠΟΛ. Άρα γιατί να ανατρέξουμε στο άρθρο 4 της απόφασης του Συμβουλίου. Αυτό δεν θα είχε κανένα νόημα. Έχει μεγάλη σημασία η νομική αποτίμηση και αξιολόγηση της Επιτροπής, όπως την ακούσαμε. Χωρίς να θέλω να πω σε άλλα ζητήματα, υπάρχουν τρεις ε, σοβαροί κίνδυνοι που ελοχεύουν μπορείτε να συμμερίζεστε τους κινδύνους ή όχι. Εγώ θα τους αναφέρω όμως για να τους σκεφτούν τα εμπλεκόμενα μέρη. Οι Βρετανοί είναι η υπέρμαχοι της εφαρμογής του 341. Λένε ότι τροποποιείται το, το πλαίσιο με βάση τη, τη δική τους την αναστολή, μάλλον την αναβολή ή διαγραφή που ζητούν. Δεν, είναι, δεν πρόκειται για Μπράμσχιλ έναντι ε, Βουδαπέστης. Μπορεί να διαγραφεί το άρθρο 4. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Δεύτερος κίνδυνος. Η Ολομέλεια μπορεί να υπερψηφίσει ή να καταψηφίσει. Αυτός είναι ένας άλλος κίνδυνος, ο οποίος δεν ε, συνυπολογίστηκε. Και ο τρίτος κίνδυνος, στον οποίο προαναφέρθηκαν μερικοί, και ο υποφαινόμενος, είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση. Δηλαδή κανονισμός που διέπει τον οργανισμό της Europol και παρεκκλήσεις με βάση τις ε, προαποφασιστήσεις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της ε, Europol. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, καταλαβαίνετε ότι τεινάζεται στον αέρα αυτή η πρόταση. Το ξέρει πολύ καλά και ο κύριος Ταβάρες. Άρα, για να είμαστε επικοδομητικοί πρόεδρε, νομίζω ότι ακολουθώντας την τακτική διαδικασία, νομική διαδικασία, θα πρέπει να φτάσουμε σε μια διαθεσμική συμφωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριο Σταβάρες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ρωτήσω κάτι την Προεδρία του Συμβουλίου. Είναι η ίδια ερώτηση που έθεσα και στον Υπουργό προλίγου. Αντιλαμβάνεστε πως ε, υπήρχε ήδη μία πρόταση της Κομισιόν και η ειλικρινή συνεργασία σημαίνει ότι κάθε όργανο της Ένωσης και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να απέχουν από δράση που θα διακινδυνεύσει έναν μια εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ αυτή εκτελείται. Πώς λοιπόν μπορεί να συμβάσετε το ότι το Συμβούλιο αποφάσισε επί νομικής πρότασης η βρίσκεται το ίδιο επιτάπητος και έχει προωθηθεί από την Κομισιόν. Πώς νομίζετε λοιπόν ότι είναι συμβατό με την αρχή της ειλικρινούς και ε, σωστής ε, συνεργασίας και δίκης συνεργασίας. Τώρα, προς την Κομισιόν. Να πω το εξής εάν η απόφαση ΣΕΠΟΛ δεν ε, τροποποιηθεί, αυτό σημαίνει ότι από νομική σκοπιά το έδρα της ΣΕΠΟΛ παραμένει στην Μπράσκουιτ. Και αυτό σημαίνει ότι το ενδιαφερόμενο κράτο μέλος δεσμεύεται να προβεί σε απαραίτητες πράξεις προκειμένου να κρατήσει την έδρα Νομίζω ότι το ερώτημα μπορεί να απαντηθεί με ένα ναι ή ένα όχι. Τρίτη ερώτηση. Τι πρέπει να κάνει τώρα το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να επικαλύψει την απόφαση, τη συναπόφαση μάλλον. Και αυτό το ερώτημα αφορά όλους μας, αλλά ίσως η νομική υπηρεσία μπορεί να μας διαφωτίσει σε τι θέση θα βρεθεί το Κοινοβούλιο από τεχνική και από πολιτική σκοπιά, εάν ακολουθήσουμε δύο άγουσες που είναι αντίθετες, αλλά Και θα ζητήσω την Προεδρία να μας απαντήσει στα όσα είπε η Κομισιόν σήμερα εδώ Όταν σου υπόθηκε ότι η απόφαση του Συμβουλίου ήταν ακατάλληλη τεχνικά και από χρονική σκοπιά ε, άσκοπη. Ευχαριστώ κύριε Αγκάτ. Ευχαριστώ. Το ίδιο ζήτημα από μια διαφορετική οπτική γωνία. Να πω πως η Κομισιόν συνεχίζει το ίδιο επιχείρημα υπέρ της συγχώνευσης. Το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ στη Λίβη και είπαμε ότι οι πολιτικές ομάδες δεν στηρίζουν αυτή την συγχώνευση. Αλλά βλέπουμε πως ε, ασκείται μία πίεση και νομίζω ότι θα πρέπει να κλείσει αυτό το θέμα της πίεσης. Τώρα, συγχώνευση ή ανεξαρτησία της ΣΕΠΟΛ και να ρωτήσω τον εισηγητή προκειμένου να μεταφερθεί από τον Πράσπη στην Βουδαπέστη. Η ερώτησή μου λοιπόν προς την Κομισιόν και στο Συμβούλιο αλλά και προς την νομική υπηρεσία έχει ως εξής ποιος θα ήταν ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προκειμένου να κλείσουμε αυτό το θέμα ασφάλεις γύρω από τα διάφορα εκκρεμή ζητήματα. Θα πρέπει λοιπόν να ολοκληρωθεί η έκθεση σχετικά με την Europol. Με τα χαράς λοιπόν θα έλεγα μια σαφή εικόνα στο τέλος της σημερινής ιστορίας για το πώς θα προχωρήσουμε και πώς θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει άλλο συνάδελφο που να έχει στήσει το λόγο, η νομική υπηρεσία. Ευχαριστώ. Σχετικά με την ερώτηση του κ. Ταβάρες. Πρώτα απ' όλα να τονίσω πως το θέμα αυτό δεν ετέθη άμεσα, αλλά μπορώ να πω ότι συνεχίζει να ισχύει η απόφαση μέχρι να ανακληθεί η πρώτη σχετικά με την ε, ΣΕΠΟΛ και όντω θα πρέπει να φροντίσει ε, η χώρα στην οποία έχει έδρα τώρα η ΣΕΠΟΛ να παρέχεται τις απαραίτητες διευκολύνσεις. Να πω ότι η συμφωνία για την έδρα της ΣΕΠΟΛ ανάμεσα, στην, ε, ανάμεσα της ΣΕΠΟΛ και την κυβέρνηση του ΙΤΑΒ, άρθρο 1 παράγραφος 3, αναφέρει ότι σε περίπτωση που τα στρατηγείο της ΣΥΠΟΛ μεταφερθεί από την επικράτεια του ΙΤΑΒ, αυτή η συμφωνία θα πάψει να ισχύει μετά από μία περίοδο που ευλόγως απαιτείται για μια τέτοια μεταφορά της ΣΕΠΟΛ. Δεν είναι λοιπόν απόλυτα ξεκάθαρο, αλλά Καταρχήν είναι προφανές πως ε, η κυβέρνηση του ΙΤΑΒ έχει την υποχρέωση να παρέχει ε, τα κτίρια και τις εγκαστάσεις της ΕΠΟΛ. Τώρα ερώτηση του κ. Ταβάρης επίσης, εάν η υπόφαση της ΕΠΟΛ τροποποιηθεί και ο κανονισμός της Europol ως προτείνει η Κομισιόν εγκριθεί, τότε ο κανονισμός της Europol θα ε, καταργήσει την τροποποιημένη απόφαση περί ΣΕΠΟΛ, αλλά μέχρι τότε μπορεί και αυτή να τροποποιηθεί με τη σειρά τη. Μπορεί να έχουμε την τροποποίηση τη απόφαση ΣΕΠΟΛ, αλλά και αργότερα μπορούμε να έχουμε με την υιοθέτηση του κανονισμού της Europol την κατάργηση της απόφασης ΣΕΠΟΛ. Αυτό είναι θέμα επιλογής του νομοθέτη. Με την έγκριση λοιπόν του κανονισμού της ε, Europol μπορεί να καταργηθεί η απόφαση περί ΣΕΠΟΛ. Τέλος υπήρχε ερώτηση από την κυρία Γκόνς νομίζω. Τι δρόμο θα ακολουθήσουμε από εδώ και μπρος. Αναφέραμε πως ε, σημασία έχει το Κοινοβούλιο να λάβει υπόψη του σύμφωνα με την κοινή δήλωση και την κοινή προσέγγιση από πολιτική σκοπιά, να λάβει υπόψη του λοιπόν τις απόψει των άλλων θεσμικών οργάνων. Αλλά αυτή η πράξη δεν είναι δεσμευτική, νομικώς δεσμευτική και μια απόφαση για τροποποίηση της απόφασης ή της κατάργησης αυτής ε, θα πρέπει να ακολουθήσει την ε, τακτική νομοθετική διαδικασία. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα βρίσκεται στα χέρια των ε, νομοθετών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η Λιθουανική Προεδρία έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Μπορώ να είμαι ιδιαίτερα σύντομος. Συμφωνώ 1000% με τα προηγούμενα σχόλια που ακούσαμε από την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου. Αυτή είναι η προσέγγιση που το, κοινο, το Συμβούλιο ακολουθούσε. Δεν είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε προηγούμενο στην υπόθεση αυτή. Τονίζω για μια ακόμα φορά ότι είμαστε, πώς να το πω, όμοιροι της υφιστάμενης κατάστασης. πως η διαδικασία της Europol έχει μπει στα σκαριά και ότι δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί έως τον Μάρτιο, γιατί αυτό είναι σαφές, και αφετέρου βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου το ΙΤΑΒ εξέφρασε την επιθυμία να λήξει να εκπνεύσει η διάρκεια της ε, έδρας τη ε, της Apple στο Μπράσχιλτ. Αυτό αναφέρθηκε πολύ σωστά από την νομική υπηρεσία. Αυτές, είναι οι πραγματικές συνθήκες. Πρέπει να δράσουμε. Συμφωνώ απόλυτα ότι θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία κυρίων ανάμεσα στα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επιληθεί το θέμα με τέτοιο τρόπο ώστε η ΣΕΠΟΛ να να μπορούν λοιπόν οι αστυνομικοί να εκπαιδεύονται καταλήλως θα πρέπει η ΣΕΠΟΛ να μπορεί να συνεχίζει τις δραστηριότητε τους. Θα πρέπει λοιπόν να λήξει αυτή η ανασφάλεια, η βεβαιότητα που ισχύει. Η Κομισιόν είπε πως έχασαν το τρένο στην θέμα, στην πρωτοβουλία του Συμβουλίου, αλλά έχουμε κάθε δυνατότητα για να προχωρήσουμε σε συμβασμού τους επικείμενες διαπραγματεύσεις, χρησιμοποιώντα ε, τις τακτικές νομοθετικές διαδικασίες. Αυτή είναι η περίπτωση και καλούμε όλα τα όργανα να κάτσουν και να βρουν την σωστή λύση, την κατάλληλη λύση. Προς το παρόν αυτή η προσωρινή λύση θα πρέπει να βρεθεί Αυτή η κοινή προσέγγιση δεν είναι νομικά δεσμευτική, αλλά δίνει το δικαίωμα στο Συμβούλιο να ορίσει το κράτος μέλος και την πόλη όπου θα εδρεύει προσωρινά αυτό, αυτή η υπηρεσία. Εάν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε αυτό το τόσο σημαντικό όργανο, υπηρεσία θα βρίσκεται σε πλήρη αβεβαιότητα και δεν ξέρω τελικά ποιος θα βγει κερδισμένος αυτή την υπόθεση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ολοκληρώσω λοιπόν τη συζήτηση για σήμερα. Κύριε Ταβάρης, παρακαλώ, ναι, επί της διαδικασίας κάτι. Ο εκπρόσωπος της Λιθουανικής Προεδρίας μας είπε ότι το κράτος μέλος είχε το δικαίωμα να ε, λήξει την ε, συμφωνία, όπως είπε και η νομική υπηρεσία. Όμως όλοι νομίζω ακούσαμε τη νομική υπηρεσία να αναφέρεται σε υποχρέωση συνέχισης με την έδρα της σε πόλη. Δηλαδή μας είπε κάτι το αντίθετο και θα ήθελα να καταγραφεί στα πρακτικά ότι η Προεδρία ρωτήθηκε για τη συμβατότητα των πράξεών της και την ε, δικαστική συνεργασία που αναφέρεται στο άρθρο 14 της συνθήκης και δεν απάντησε. Θα θέλατε να αντιδράσετε σε αυτό. Ναι, επαναλαμβάνω. Ούτε και το Συμβούλιο προτιμά μια τέτοια κατάσταση. Δεν μας αρέσει η κατάσταση του Ηνωμένου Βασίλειου να λύγει μια συμφωνία, να κυρώνει μια συμφωνία. Υπήρξε όμως μια συμφωνία να σταματήσει η Σεπόλ να εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο και αυτό ήταν βάση για περαιτέρω αναλύσεις. Και ίσως όλα τα θεσμικά όργανα θα έπρεπε να λάβουν υπόψη γνωμοδοτήσεις των νομικών υπηρεσιών σχετικά με κυρώσεις, πιθανές κυρώσεις οι οποίες θα μπορούσαν να επιβληθούν εδώ και πάλι να πω ότι είναι θέμα διαπραγματεύσεων οι συνέπειες της ε, λύσης αυτής ε, της σχέσης για την έδρα της ΕΠΟΛ. Και αυτή είναι μια πρωτοβουλία που ανέλαβε το Συμβούλιο και να τονίσω ότι από τα 25 κράτη-μέλη, ε, ξέρετε η Δανία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί έχουν διαφορετικό καθεστώς. Σας ευχαριστώ. Θα θέλετε να παρέμβετε. Ναι, σύντομα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε την ευκαιρία να πει την τελευταία φορά ενώπιον της Επιτροπής αυτή την αποψή της. Από τότε μέχρι τώρα έχουμε σημειώσει πρόοδο. Να σας πω ότι σημειώσαμε την επικοδομητική πρόοδο που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στους δύο αυτούς συνομοθέτες για αυτή την νομοθετική πρόταση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να στηρίξει και να συνεχίσει αυτήν την καλή συνεργασία και καλή πρόοδο. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ζήτημα της έδρας της ΕΠΟΛ πρέπει να εξεταστεί στα πλαίσια της ε, λειτουργικής και επιχειρησιακής μεταρρύθμισης της ε, δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας. Η Επίτροπος επιμένει στην ε, συγχώνευση και είναι ξεκάθαρο ότι μετά από πολλούς μήνες συζητήσεων και διαπραγματεύσεων ότι εμείς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είμαστε ανοιχτοί στην εξέταση κάθε πιθανού ενδεχομένου, κάθε πιθανού διακανονισμού, ενός διακανονισμού όμως ο οποίος θα σέβεται τις συνέργειες και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί. Και εδώ να πω ότι καλωσορίζω την πρόταση του εισηγητή κ. Ντίας Δεμέρια να υπάρξει μια διοργανική συμφωνία ή έστω μια διοργανική συζήτηση κατά την οποία θα εξετάσουμε νέες επιλογές. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο μιας ε, συστέγασης σε Πολ και Ευρωπόλ, διατηρώντας όμως παράλληλα την ανεξαρτησία των δύο αυτών οργανισμών, καθώς και την ε, λειτουργική και επιχειρησιακή αυτονομία τους. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θέλουμε να εκφράσουμε την ανησυχία μας για την ΕΣΕΠΟΛ και για το προσωπικό της ΕΠΟΛ και θα εκτιμήσουμε οποιαδήποτε διασφάλιση μπορεί να δοθεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνουμε λοιπόν με εσάς το σημείο αυτό της ημερησίας διάταξης. Ευχαριστώ πολύ όλους όσους συμμετείχαν στη συζήτηση. Πιστεύω πως δεν έληξε εδώ το θέμα αυτό. Ας προχωρήσουμε τώρα στο σημείο 7 της ημερησίας διάταξης, την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα. Για το 2011 μέχρι το 2013 η συγγήτρια είναι η κυρία Ιντφέλτ. Εάν θυμάστε, η έκθεση αυτή προβλέπεται από το άρθρο 104 του εσωτερικού κανονισμού. Και, και στο παρελθόν έχουν ήδη παρουσιαστεί δύο σχετικές εκθέσεις. Η τελευταία ήταν η έκθεση Χάουταλα Αργεντίνη. Δεν θα μπω όμως σε λεπτομέρειες. Θα δώσω κατευθείαν στο, τον λόγο στην κυρία Ιντφέλτ να προσθέσω μόνο ότι... Συνάδελφοι, παρακαλώ εγκαταλείψτε την αίθουσα αν επιθυμείτε, αλλά χωρίς θόρυβο. Yes, I need to be more strict. So, uh, we were informed that uh, Mrs. Sommer will be replaced. Ο κύριος Φως θα αντικαταστήσει την κυρία Ζόμερ, ο σκιώδης εισηγητής του ΑΕΛ και η κυρία Ιντφέιντ Τώρα έχει το λόγο και μετά οι σκιώδεις εισηγητές. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Πράγματι, χρειάστηκε καιρός για να μπει πάλι στην ημερήσια διάταξη έκθεση αυτή μετά τις εκθέσεις Χαουταλά και Σαρτζεντίνη. Και πιστεύω πως ε, θα ακολουθήσει μια πολύ σοβαρή συζήτηση για το ζήτημα της διαφάνειας και της πρόσφασης στα έγγραφα, κάτι που προσωπικά πιστεύω είναι κέριο για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν κοιτάξουμε το παρελθόν και τα παρασκήνια αυτής της έκθεσης, συνειδητοποιούμε καταρχάς ότι τώρα πλέον έχει τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας και δεύτερον υπάρχει νέα νομολογία από τότε που δημοσιεύτηκε η τελευταία έκθεση. Και οι αλλαγές αυτές έχουν επέλθει από προτάσεις που εγώ ίδια υπέβαλα. Δεύτερον, Πιστεύω πως δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το γεγονός ότι οι πολίτες ζητούν έντονα περισσότερη διαφάνεια, ζητούν πρόσβαση στα έγγραφα. Πολύ συχνά το Συμβούλιο και η Κομισιόν, ιδιαίτερα το Συμβούλιο, επιχειρηματολογούν λέγοντας ότι η περισσότερη διαφάνεια ενδεχομένως βλάψει ορισμένες ε, διεθνείς διαπραγματεύσεις, για παράδειγμα. Και πιστεύω πως η άκτα, η συμφωνία άκτα έδειξε πως το αντίθετο ισχύει, πως η έλλειψη διαφάνειας βλάπτει τις διαπραγματεύσεις. Και γιατί αυτό, γιατί οι πολίτες χάνουν την εμπιστοσύνη τους. Και για μένα το κεντρικό σημείο της συζήτησης είναι το πώς θα αλλάξουμε την παλιά διπλωματική κουλτούρα όπου οι διπλωμάτες και οι δημόσιοι υπάλληλοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο και όλα διενεργούνταν κάτω από απόλυτη μυστικοπάθεια και χεμήθεια. Πώς θα αλλάξουμε λοιπόν την ε, κουλτούρα αυτή και θα την κάνουμε πιο ανοιχτή έτσι ώστε να προσαρμοστεί σε μια απόλυτα δημοκρατική Ευρώπη των πολιτών η οποία ένωση και οι πολιτική θα λογοδοτούν. Έχει λοιπόν ε, τη στήριξη της κοινή γνώμης η πρόταση αυτή. Η έκθεση τώρα δεν είναι πολύ μεγάλη, καταρχάς σε κάτι τεχνικό. Καθώς συνέτασα την έκθεση αυτή, και να σας πω ότι είχα βιαστεί να το κάνω, δεν είχα πολύ χρόνο, οι προτάσεις μου κατέληξαν στις αιτιολογικές σκέψεις παρά στα άρθρα καθ' αυτά και αυτό θα το διορθώσω με τροπολογίες. Αυτό ιδιαίτερα ε, έχει σχέση με τα σημεία και, A T. Δεν θέλω να επαναλάβω όλες τις ε, συστάσεις οι οποίες ήταν εξαιρετικές ε, στις έκθεσεις ε, Σαρτζεντίνη και Χαουτάλια. να πω ότι λείπουν κάποιες από αυτές, όμως θα συμπεριληφθούν και γι' αυτό θα ήθελα το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιδράσουν και να απαντήσουν στις συστάσεις αυτές. Και αυτή είναι την σύσταση κάνω εγώ προσωπικά, ότι πρέπει να υπάρχουν αιτήσιες εκθέσεις σχετικά με την διαφάνεια και την πρόσβαση στα έγγραφα. Προτείνω λοιπόν να αντιδράσουν μέσω της αιτήσιας εκθεσής τους στις προτάσεις του Κοινοβουλίου. Η δεύτερη σημαντική σύσταση, που είναι και αυτονόητη, πιστεύω, είναι ότι εμείς θεωρούμε επίγον να δημιουργηθεί ένας ε, αναθεωρημένος κανονισμός. Είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, αυτό το μπλοκάρισμα και πιστεύω πως πρέπει να λυθεί το θέμα άμεσα. Ορισμένοι συνάδελφοι άκουσα πως πρότειναν απλά να καταπιούμε έτσι αμάσιτες τις προτάσεις της Κομισιόν για λιγότερη διαφάδη, μια έτσι για να τελειώσουμε πριν λήξει και η θητεία μας. Εγώ ποτέ δεν πρόκειται να στήριξω μια τέτοια πρόταση. Το οφείλουμε στους πολίτες μας να πολεμήσουμε μέχρι το τέλος για περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη λογοδοσία και όχι λιγότερη. Επίσης, επιχειρηματολογώ υπέρ απλουστευμένων διαδικασιών. Έχω πολλή εμπειρία προσωπικά όσον αφορά την ε, αίτηση για έγγραφα. Όταν μου αρνείται η πρόσβαση σε έγγραφα, η μόνη οδός και ο μόνος τρόπος που έχω για να ε, ε, τα αποκτήσω είναι να προσφύγω στο δικαστήριο και κάτι τέτοιο απαιτεί χρόνια. Για μια τέτοια περίπτωση βρίσκομαι πέντε χρόνια στα δικαστήρια και δεν προβλέπεται ημερομηνία καταληκτική και το κόστος είναι απαγορευτικό μιας τέτοιας διαδικασίας. Εμείς λοιπόν θα θέλαμε μια απλουστευμένη διαδικασία, πολύ απλουστευμένη. Εδώ προτείνεται να καταφεύγουμε και να προσφεύγουμε στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, που πιστεύω πως είναι μια πολύ τιμή πρόταση. Ωστόσο, δεν μπορούμε να ε, αναγκάσουμε τον Διαμεσολαβητή να δράσει γρήγορα και να αποφανθεί γρήγορα. Χρειάζομαστε λοιπόν περισσότερες ε, και μη επαχθείς διαδικασίες, έτσι ώστε να μειωθεί η δικαστική γραφειοκρατία. Επίσης, κάτι που προτείνω και πιστεύω ότι θα μπορούσαν να κάνουν ήδη από χθε τα θεσμικά όργανα, είναι η διαφάνεια, είναι να δημιουργηθεί ε, μια υπηρεσία διαφάνειας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν ε, ε, στις, σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες γραφεία έχει θα μπορούσαμε να αλλάξουμε τα δεδομένα και να ορίσουμε έναν υπεύθυνο διαφάνειας. Έπειτα, προτείνω όλα τα θεσμικά όργανα και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναθεωρήσουν τους εσωτερικούς κανονισμούς τους όσον αφορά την καταγγελία παρατυπιών. Η καταγγελία παρατυπιών δεν θα πρέπει να αποκλείεται ως ένα από τα μέσα της πρόθεσης της διαφάνειας, ως ένα από τα δημοκρατικά μέσα πρόθεσης της διαφάνειας. Και πιστεύω πως ε, πρέπει πρώτα να αναθεωρήσουμε τους εσωτερικούς μας κανονισμούς για την καταγγελία παρατυπιών και να φροντίσουμε έτσι ώστε όσοι τις καταγγέλουν να απολαμβάνουν τις ε, καλύτερες δυνατές προστασίες. Στην ετήσια επίση έκθεση του Συμβουλίου και της Κομισιόν για την διαφάνεια θα πρότεινα να βελτιωθεί η διαμόρφωση έτσι ώστε να μπορούμε να συγκρίνουμε πολύ πιο εύκολα τα στατιστικά στοιχεία. Μετά, υπάρχει ένα σχόλιο για την, τα προγράμματα επιοίκειας και υπάρχει τώρα μια πρόταση, μια πίεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία μιας, ε, ενός συστήματος αυτόματης εξαίρεσης από τους κανόνες διαφάνειας για προγράμματα επίοικειας. Ε, δεν θα πω σε λεπτομέρειες γιατί είναι εξαιρετικά τεχνικό το θέμα αυτό, απλώς ήθελα να το αναφέρω και να πω, ολοκληρώνοντας, ότι χρειάζεται να δούμε την τυπική εφαρμογή των ε, λόγων εξαίρεσης από την ε, Κομισιόν και το Συμβούλιο. Ιδιαίτερα την εξαίρεση για την προστασία των διεθνών σχέσεων. Αυτό είναι κάτι που χρησιμοποιούνται συνέχεια, είναι πλέον ρουτίνα και γίνεται υπερβολική χρήση του. Και στην ε, νομολογία αυτό χρησιμοποιείται συνεχώ και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το Συμβούλιο και η Κομισιόν αρνούνται να εφαρμόσουν τι αποφάσει του δικαστηρίου. Τέλο. Χρειαζόμαστε διαδικασίε, χρειαζόμαστε κριτήρια, χρειαζόμαστε ε, κανόνε για την ε, διαβάθμιση των εγγράφων, διότι έχουμε μεν τον κανόνα για την διαφάνεια, όμως, εάν το Συμβούλιο, η Κομισιόν, το Κοινοβούλιο, η Ευρωπόλη, οποιοδήποτε άλλος αποφασίσει να ε, χαρακτηρίσει, να ταξινομήσει ένα έγγραφο ως ε, απόρριτο, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να προσφύγεις στο δικαστήριο, δεν υπάρχει κανένας ε, κανόνας για το πώς χαρακτηρίζεται ένα έγγραφο. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις που θα θέτουν κριτήρια και προϋποθέσεις για αυτό. Και χρειαζόμαστε επίσης ένα εποπτικό σώμα, το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τέλος, να πω ότι ως εισηγήτρια έχω κάθε πρόθεση να δω με πολύ κριτικό και επικριτικό βλέμμα της πράξης του Κοινοβουλίου. Και να πω ότι δεν πρέπει να μένουμε στα λόγια και θα έπρεπε να, να ιδρύσουμε και εδώ ένα γραφείο διαφάνειας. Τέλος, να πω ότι προθεσμία υποβολής τροπολογιών 13η Ιανουαρίου. Σκοπεύουμε να ψηφίσουμε στην Επιτροπή Λίμπε τον Φεβρουάριο και μάλλον στην Ολομέλεια του Μαρτίου, γιατί πιστεύω πως δεν θα προλάβουμε στην δεύτερη Ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Αυτά προς το παρόν. Θα χαρώ πολύ να ακούσω τα σχόλιά σας και να λάβω τις τροπολογίες σας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Εφός θα λάβει το λόγο ως αντικαταστάτης της κυρία Ζόμερ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. να σας πω δυστυχώ ότι πρέπει να ψηφίσω σε μια άλλη επιτροπή και δεν θα καταφέρω να ακούσω την απάντησή σας. Θα ήθελα όμως να τοποθετηθώ εκ μέρους της κυρίας Ζόμερ που πρέπει να απουσιάσει δυστυχώ το ΕΛΚ. Υποστηρίζουμε την αρχή της περισσότερης διαφάνειας. Όσο περισσότερη τόσο το καλύτερο. Διερωτώμαστε απλά εάν η υπερβολική διαφάνεια οδηγήσει σε αδιαφάνεια, γιατί όταν υπάρχει ένας κατακλυσμός πληροφοριών, υπάρχει και σύγχυση και δεν μπορούμε να βρούμε ακριβώς αυτό που θέλουμε. Γι' αυτό πιστεύω πως θα έπρεπε να βρούμε την σωστή ισορροπία, το πώς ακριβώς ε, θα έχουμε πρόσβαση σε έγγραφα, πόση, πώς ακριβώς θα είναι διαρθρωμένη η διαφάνεια διότι πραγματικά πιστεύω ότι όταν δημοσιεύονται τα πάντα υπάρχουν και πολλά ασήμαντα στοιχεία που μπερδεύουν. Τώρα, όσον αφορά την διαδικασία και για τα ουσιώδη και τα μη ουσιώδη, να πω ότι ο κανονισμός του 2009 είναι πλέον παλιός και πρέπει να επικαιροποιηθεί, να επικαιροποιηθεί και σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Εγώ προτείνω να, η κυρία Σόμερ μάλλον προτείνει να υπάρξει δυνατότητα προσαρμογής, επικαιροποίησης, όπως και με, τους αντίστοιχους, με τις αντίστοιχες περιπτώσεις του 2011. Αλλά σε αυτήν την περίπτωση θα μπορούσαμε να εστιάσουμε σε αυτό που είναι πρακτικό, εφικτό και συνετό και να μην προσφέρουμε στους πολίτες τα πάντα, αλλά τα ουσιώδη, αυτά που χρειάζονται. Τώρα, κάτι που προσωπικά ήθελα να τονίσω είναι τα έγγραφα διαπραγματεύσεων, διεθνών διαπραγματεύσεων. Η άκτα που αναφέρατε ήταν ένα παράδειγμα κατά το οποίο δεν υπήρξε απόλυτη διαφάνεια. Έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά το περιεχόμενο είχε να κάνει με τον περιορισμό της ελευθερίας στο διαδίκτυο. Τώρα, εάν ε, η εξέλιξη και τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων της ΑΚΤΑ είχαν άμεση σχέση με την διαφάνεια ή την έλλειψη αυτή, είναι κάτι για το οποίο δεν είμαι σίγουρος. Αλλά σίγουρα εμείς μπορούμε να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες. Όμως όσον αφορά την διαπραγματευτική μας θέση κατά τη διάρκεια διεθνών διαπραγματεύσεων ε, δεν είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι θα βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων μας, αν θέλουμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και πιστεύω πως συνεδριάσεις μας μεταδίδονται μεν, αλλά όχι όλες τις φορές. Κάποιες συνεδριάσεις γίνονται και κλεισμένων των θυρών, διότι πρέπει να συζητηθούν κάποια ε, θέματα που έχουν σχέση με τις ε, διαπραγματεύσεις, με την ε, θέση μας. Και δεν θα ήθελα εγώ προσωπικά να είναι ενημερωμένος ο... Ε, αντίπαλος εντό αγωγικών σε μια διαπραγμάτευση για το ποια στρατηγική θέλω να ακολουθήσω. Τώρα πιστεύω πως σε γενικές γραμμές η πρόταση είναι καλή. Η αξία όμως που δίνω εγώ, η δική αξία, είναι στις συστάσεις και την εφαρμογή τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εφαρμογή όμως των συστάσεων αυτών πρέπει να είναι καλυμμένη από μια σωστή νομική βάση. Όταν έχουμε την κατάλληλη νομική βάση πιστεύω πως θα μπορούμε και να την εφαρμόσουμε. Εάν λείπει, τότε θα έχουμε δυσκολίες. Πρέπει να υπάρχει νομική βάση για την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουμε και αν δεν την έχουμε τότε δυστυχώς χάσαμε, πρέπει να τη δημιουργήσουμε. Χωρίς νομική βάση όμως δεν πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Τώρα, σε γενικές γραμμές, να πω κάτι σχετικά με τη διαδικασία. Η συγγήτρια το ανέφερε ήδη και πιστεύω πως είναι μια πολύ καλή ιδέα. Θα μπορούσαμε ίσως να την ε, σταχυολογήσουμε κάπως. Πολλές φορές διαβάζοντας το κείμενο έχω την αίσθηση ότι όταν μιλάει για κάποιον ε, ειδικό, για κάποιο γραφείο διαφάνειας, έχω την αίσθηση ότι κάπως ε, συγχέονται τα πράγματα. Πρέπει και συμφωνώ να βρεθεί κατάλληλη υποδομή, αλλά πιστεύω πως ε, δεν πρέπει να περιπλέξουμε τα πράγματα. Εφόσον υπάρχει μία νομική διαδικασία, πρέπει καταρχάς να καταστεί αυτή σαφέστερη, έτσι ώστε να δούμε ποιες νομικές δυνατότητες έχουμε και πώς αυτές μπορούμε να τις εφαρμόσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε γενικές γραμμές ε, όμως, εμείς ως ΕΛΚ επιθυμούμε μία λιγότερο γραφειοκρατική διοίκηση. Γι' αυτό και πιστεύω πως οι προτάσεις που αναφέρονται σε αυτό είναι σωστές. Χρειάζονται αυτές οι ελαφριές υποδομές. Τώρα, το αίτημα για περισσότερη διαφάνεια και η κοινή γνώμη, να πω ότι υπάρχουν ορισμένα φόρουμ που το ζητούν, όχι η πλειοψηφία των, ε, της κοινή γνώμης και λαμβάνοντας υπόψη και τις πρόσφατες γερμανικές εκλογές, δεν μπήκαν στο Γερμανικό Κοινοβούλιο όλοι όσοι ζητούσαν την απόλυτη διαφάνεια. Οπότε για τη δική μου χώρα τουλάχιστον δεν μπορώ να πω ότι αυτό φαίνεται απόλυτα και από την ε, κοινή γνώμη. Υπάρχει όμως ένα κίνημα, σίγουρα, και υπάρχει επίσης σίγουρα ένα μεγάλο ενδιαφέρον για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το παρελθόν ε, μιας πράξης, μιας διαπραγμάτευσης, αλλά δεν θα έλεγα ότι η κοινή γνώμη είναι απόδειξη της ε, μεγάλης ανάγκης για περισσότερη πληροφόρηση, περισσότερη γνώση. Εδώ θα έλεγα ότι δεν είναι για μένα κάτι που θα έχει ως επακόλουθο την αλλαγή. Είναι κάτι που υπάρχει γενικά, είναι μια τάση που υπάρχει στην κοινωνία, όχι απέτηση. Γι' αυτό λοιπόν θα προτείνω ορισμένε μικρέ τροποποιήσει, βελτιώσεις έτσι ώστε ε, το αίτημα για διαφάνεια να γίνει πιο ξεκάθαρο και πιο στοχευμένο και να μην ε, πνιγεί από υπερβολικές πληροφορίες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φώση, κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ την κυρία Ιντβέλτ για την εξαιρετική αυτή έκθεση, την άκρος ενδιαφέρουσα. Δεν είναι συνέχεια της έκθεσης Χάουταλα, δεν την αντιμετωπίζω εγώ έτσι, είναι ε, επιβεβαίωση της εργασίας του ε, Μάικλ Κάσμεν για την ελεύθερη πρόσβαση σε δημοσία έγγραφα. Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι εμεί που ζητούσαμε περισσότερη διαφάνεια προσπαθούμε να βρούμε και λύσεις σε ένα τόσο περιορισμένο τομέα. Δηλαδή εσείς ε, μιλάτε για ένα γραφείο διαφάνειας αναθεσμικό όργανο. Αλλά σε αυτή την περίπτωση θέλουμε να υπάρχει μία κοινή διαχείριση χωρίς να υπάρχει το, τόση εχεμήθεια ή μυστικοπάθεια στη χειρότερη περίπτωση. Θα ήθελα λοιπόν να συνεργαστούμε και με τον εισηγητή ε, μιλώντας για δημοσιοποίηση των εγγράφων, εκτός και αν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για λόγους δημόσιας τάξης ή ασφάλειας. Ε, πέρσι συζητήσαμε ένα εγγραφό της Επιτροπής Προπολογισμών σε σχέση με τον διερευνητικό ε, διερευνητική δημοσιογραφία. Αυτή ήταν μια πολύ καλή πρωτοβουλία. Δεν πρέπει όμως να τα περιορίζουμε όλα αυτά για να μην έχουμε περιθώρια δράσης. Αναφερθήκατε στην άκτα και θυμάμαι και τις διαπραγματεύσεις με τις ΙΠΑ. Υπάρχει έλλειψη διαφάνειας ως προς τις διαπραγματεύσεις αυτές δεν ε, χρειάζεται να ε, δημοσιοποιήσετε την στρατηγική σας, αλλά θα πρέπει να είσαστε ανοιχτοί με τους πολίτες. Αυτό που με εκπλήσει σε αυτή την προσέγγιση όπου όλα είναι απορρίτου χαρακτήρα εκτός και αν, υπάρχει αυτό το εκτός και αν, ε, ε, είναι ότι κινούμαστε προς μια προεκλογική εκστρατεία όπου οι πολίτες εμπιστεύονται τους πολιτικούς όλο ένα, και λιγότερο. Κάνουμε λάθη, αλλά θα πρέπει οι πολίτες να μπορούν να παρακολουθούν τις εργασίες μας. Ξέρουμε ότι το σφάλμα είναι κάτι το ανθρώπινο θα πρέπει να βρούμε και άλλες λύσεις. Ο Ombudsman να έχει περισσότερα περιθώρια ε, διερεύνησης ή έρευνας, οι δημοσιογράφοι να έχουν μεγαλύτερα περιθώρια ελιγμών και να μπορούμε να ακούμε καλύτερα και τους καταγγέλλοντες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ. Θα μιλήσω αγγλικά αυτή τη φορά. Ευχαριστούμε για την εξαιρετική αυτή έκθεση, την εισηγήτρια. Αυτά ακριβώς περιμέναμε από τη Σοφή Ιντβελτ. Όπως είπε και η κυρία Σαρτζεντίνη, λυπάμαι γιατί λίγους μήνες πριν από τις ευρωεκλογές ε, υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται και δεν θέλουν πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πείρα μου είναι διαφορετική. Ε, υπάρχει έλλειψη γνώσης, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν την αποζητούν οι πολίτες. Οι πολίτες θέλουν ε, πολύ περισσότερα. Μιλάμε για την TTIP με τις ΗΠΑ, τη νέα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και εκτός από ορισμένες διαρροές δεν γίνεται ε, μια δημόσια συζήτηση για μια τόσο σημαντική συμφωνία με τις ΗΠΑ. Θα ήθελα να υπάρξει πλήρης διαφάνεια και εάν υπάρχουν θέματα τεχνικής υφής που δεν πρέπει να αποκαλύψουμε, τουλάχιστον ας ε, πούμε στους πολίτες τι διαπραγματευόμαστε. Επίσης μιλάμε για ανοιχτό χαρακτήρα των τριμερών διαλόγων γιατί σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν διαπραγματευτές ε, με ανοιχτές διαπραγματεύσεις, ενώ εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλα γίνονται και κλεισμένων των θυρών. Θα πρέπει να πούμε στο Συμβούλιο ότι αυτά είναι τα, αυτές είναι οι προδιαγραφές μας, υπάρχει διαφάνεια, αλλά δεχόμαστε τις θέσεις του Συμβουλίου για τέτοιες διαπραγματεύσεις. σε ορισμένους τομείς νομίζω ότι είμαστε ε, πολύ ευγενείς. Λυπάμαι που δεν έχει επιτελεστεί πρόοδος για το 1049 και την αναθεώρηση αυτού του κανονισμού του 2001. Νομίζω ότι μπορούμε να ε, ε, χρησιμοποιήσουμε πιο έντονη γλώσσα και αυτό μπορεί να γίνει κατανοητό το Κοινοβούλιο έχει προβάλει μια θέση στην ομάδα εμπειρογνωμόνων. Είναι πολύ καλό αυτό που αναφέρατε, δηλαδή την πρόσφατη πρόοδο που έχει επιτελεστεί ως προς τους καταγγέλλοντες. Νομίζω ότι η σύσταση δεν είναι ε, σαφής. Νομίζω ότι θα πρέπει να πιέσουμε εδώ. Αυτά θα ήθελα να πω. Ε, χαίρομαι για το σχέδιο έκθεσης και δεν θα ήθελα να αποδυναμωθεί. Ευχαριστούμε κύριε Νταϊόν ή Σοφή. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω στα Ολλανδικά. Συνήθως δεν το κάνω, αλλά αυτή τη φορά θα κάνω μία εξαίρεση. Το ΕΛΚ δεν είναι πια παρόν, γι' αυτό ίσως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και ορισμένα ε, άλλα στοιχεία. Υπάρχει η πρόταση υπερβολική διαφάνεια. Δεν το κατανοώ αυτό. Πώς μπορεί να υπάρχει υπερβολική διαφάνεια. Υπάρχουν χώρες όπου η πληροφορία, οι πληροφορίες μπαίνουν στο διαδίκτυο, εκτός και αν υπάρχει σοβαρός λόγος για να μην γίνει κάτι τέτοιο ως προς τον απόρριτο χαρακτήρα στον, στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, δεν χρειάζεται να επανεφεύρουμε το τροχό. Το ΕΛΚ ε, γνωρίζει ότι υπάρχει νομολογία επί του θέματος. Δικηγόροι και δικαστές ε, οι οποίοι λένε τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν μπορούμε αυτόματα να κάνουμε να μετατρέπουμε τα στοιχεία σε απόρριτα. Θα πρέπει να έχουμε μία στρατηγική προσέγγιση. Δηλαδή υπάρχουν στοιχεία απορρίτου, αλλά όχι ολόκληρο το κείμενο. Αυτό θα πρέπει να αιτιολογηθεί και αυτό μας δείχνει και η νομολογία. Ως προς την σύσταση νέων ε, θεσμών, ή οργανισμών. Δεν θέλω να συσταθούν ε, νέοι οργανισμοί. Και αυτό το λέω προς την κυρία Σαρτζεντίνη ιδιαίτερα. Θα πρέπει να υπάρχει δημόσια πρόσβαση στους ε, κανονισμούς και στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Ακόμα όμως και αν υπάρχει θέληση για κάτι τέτοιο δεν σημαίνει ότι είναι λειτουργικό έμπρακτα. Υπάρχει και η διαδικασία ταξινόμησης και επιμερισμού του απορρίτου. Δεν υπάρχει κανένα καθεστώς αποπτίας. Εάν υπάρχει μία αρνητική απόφαση, ε, πρέπει κανείς να προσφύγει στις δικαστικές αρχές. Αυτό είναι ιδιαίτερα, φορτώνει ιδιαίτερα την όλη διαδικασία. Ως προς τον ε, επόπτη διαφάνειας δεν μπορώ να τον φανταστώ να λαμβάνει υπόψη, δηλαδή ε, υπόψη με μονομένες αναφορές όπως είπε ο κύριος Φως. Είναι κάποιος που συμβουλεύει. Θα υπάρχει μια ετήσια ε, έκθεση για το μη απόρριτο ή την άρση του απορρίτου ή τη διαφάνεια. δηλαδή μία μερόληπτη προσέγγιση των πραγμάτων. Προσβλέπω τις τροπολογίες από τους πράσινους και την ΚΟΕ για να προωθηθεί ε, περισσότερο αυτή η έκθεση, να ενδυναμωθεί, να ενισχυθεί. Και έγινε λόγος και για τις ευρωεκλογές, αυτή τη συνάφεια με τις ευρωεκλογές. Εάν ε, θέλετε να παραμείνετε στο σκοτάδι, ψηφίστε ΕΛΚ. Αν θέλετε ανοιχτή δημόσια διοίκηση, ψηφίστε κάποιον άλλον. Αυτό είναι το μανιφέστο. Μέχρι τις εκλογές δηλαδή. Έχουμε τις εκκρεμούσες ε, διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση των κανονισμών. Τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να δείξουν ποια είναι η θέση τους. Αυτό είναι ο κατάλληλο χρόνος και σε αντίθεση με αυτά που είπε ο κύριο Φω, νομίζω ότι ενδιαφέρονται οι άνθρωποι. Ενδιαφέρονται οι πολίτες. Μπορείτε να σκεφτείτε ό,τι θέλετε για το ε, Wikileaks, για το Anonymous, σκεφτείτε ό,τι θέλετε. Οι άνθρωποι όμως θέλουν να ξέρουν. Δηλαδή θα πρέπει να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν οι άνθρωποι επιλέξουν να μην θέλουν τη γνώση, είναι δική τους επιλογή. Αλλά νομίζω ότι γενικά ενδιαφέρονται και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο στην προεκλογική εκστρατεία. Ευχαριστούμε κυρία Ιντφέλτ. Αν δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο, πάμε στο επόμενο θέμα. Μιλήσατε για τις ε, προθεσμίες, ναι, 13 Ιανουαρίου είναι η προθεσμία υποβολής ε, τροπολογιών. Ωραία. Είναι η προθεσμία λοιπόν 13 Ιανουαρίου. Τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ε, εκτίμηση της δικαιοσύνης στον τομέα της ποινική δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου. Δίνω το λόγο στην κυρία Γκέντς που θα μας παρουσιάσει την έκθεσή της Ζητήθηκε άδεια για την έκθεση, για την ε, σύνταξη αυτής της έκθεσης. Στις 27 Νοεμβρίου εδόθη η άδεια και τώρα περιμένουμε την ε, τελευταία απόφαση από την διάσκεψη των Πρόεδρων. Κύριε Αγγέντς. Να ξεκινήσω λοιπόν με τα διαδικαστικά. Περιμένουμε λοιπόν την τελική άδεια από το Μάιο, πάνω από έξι μήνες δηλαδή. Τότε οι συντονιστές ομοφόνος ενέκριναν την ε, έκθεση και υπήρξε μια διαμάχη με την Γιούρε αναφορικά με τον τίτλο και το πεδίο της έκθεσης ε, και τον Νοέμβριο στη διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών θεωρήσαμε ότι θα ληφθεί μια απόφαση από το Προεδρείο την περασμένη εβδομάδα, αλλά ακόμα την περιμένουμε, αυτή την έγκριση. Καταρχήν να σας ρωτήσω ως πρόεδρος της σημερινής μας συνεδρίασης να ζητήσετε από την διάσκεψη των Προέδρων να το θέσουν στην επόμενη μισή διάταξη της συνεδριάσεώς τους, διότι δεν να περιμένουμε άλλο. Και γνωριζόμαστε ότι χρειάζεται κάποιους χρόνους για τις μεταφράσεις. Και από ό,τι γνωρίζω, οι περισσότερες ομάδες έχουν ορίσει και σκιώδεις ηγητές, εκτός από το ΕΛΚ νομίζω. Λοιπόν, επειδή είναι πήγον το θέμα, παρακαλώ προβείτε στο απαραίτητο διάβημα προς τη διάσκεψη των Προέδρων. Τώρα, σχετικά με το περιεχόμενο, να υπενθυμίσω πώς ξεκίνησε το θέμα. Όταν η Επιτροπή λοιπόν παρουσίασε την ανακοίνωσή της για τον πίνακα του δικαιοσύνης ε, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα θέματα ποινική δικαιοσύνης ε, και τα ε, θέματα κράτους δικαίου γιατί είναι σημαντικά και επίσης οι συνθήκες παρέχουν την απαραίτητη νομική βάση για όλα αυτά τα ζητήματα κράτους δικαίου, ποινική δικαιοσύνη κλπ. Επίσης και το ζήτημα της ανεξαρτησίας δικαιοσύνης είναι ένα θέμα που τίθεται για κάποια κράτη και με αυτό θα ασχοληθεί η έκθεσή μου. Σημασία για μας έχει επίσης να μπορείς να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατόν με την αξιολόγηση του κράτους δικαίου στα κράτη-μέλη. Σήμερα συζητήσαμε το θέμα κατά τη της παρουσίας της κυρίας Ρέντινγκ εδώ για την περαιτέρω ενίσχυση των μηχανισμών για τήρηση του άρθρου 2 για των θεμελιδών αρχών της Ένωσης. Επίσης είχαμε διάφορες συζητήσεις να γίνονται όλα σε ισότιμη βάση, να αποφεύγουμε ε, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Στην έκκληση αφενό λέμε ότι ο πίνακα ο σχετικός με τη δικαιοσύνη θα πρέπει να αφορά όλες τις πτυχές συμπεριλαμβάνει τη ε, ποινική ε, δικαιοσύνη ε, την ανεξαρτησία των δικαστήριων και των δικαστών και το επίσης σήμερα ακούσαμε την κυρία Ρέντινγκ ότι υπήρξαν κάποιες δυσκολίες φέτος ελπίζω να μην έχουμε τα ίδια προβλήματα και φέτος Το scoreboard θα πρέπει να υποβάλλεται και στα εθνικά κοινοβούλια. Να υπάρχει δηλαδή ανάμειξη των κοινοβουλίων, των εθνικών. Και ζητάμε επίσης ένα μηχανισμό για αξιολόγηση της συμμόρφωσης σχετικά με τις θεμελιώδεις αρχίες που <coughs> περιγράφονται στην συνθήκη. Στην αρχή ζητήσαμε την Επίτροπο κυρία Ρέντινγκ πότε θα μας τα παράσει όλα αυτά η Κομισιόν. Ελπίζω να μην προκαλέσουμε διαμάχες όπως αυτή με τη ΣΕΠΟΛ. Χρειάζεται λοιπόν ε, να κάνουμε κάτι ώστε η διάσκεψη των Προέδρων να μας δώσει επιτέλους την άδεια να προχωρήσουμε σε αυτό το τόσο σημαντικό και επίγον θέμα. Επειδή υπάρχει μόνο ένα μέλος ανάμεσά μας, ε, ό,τι φαίνεται δεν θα αναλάβει το λόγο. Κατάλαβα λοιπόν αυτά τα οποία είπατε. Θα ζητήσω την γραμματεία να προετοιμάσει μια επιστολή. Αλλά έχουμε όμως ήδη ημερομηνία κάθε τροπολογιών. Παράξενο είναι αυτό. Α, όχι. Δεν θα αναβληθεί αυτή η προθεσμία, θα μετατεθεί η προθεσμία που είχαμε θέσει για τροπολογίες. Ευχαριστώ λοιπόν όλους και όλες ε, που μείνατε μέχρι το πέρας της συνεδριάσεως. Κλείνουμε τώρα τη συνεδρία, θα ξεκινήσουμε αύριο το πρωί στις 9. Ευχαριστώ, καλό βράδυ.